because we will finish at 10 at 3. Colleagues, please, I ask you to... Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Dear colleagues, Ε, ε, ε. Please, let's start. Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι να ξεκινήσουμε. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο στη μερίσια διάταξη και πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τις 10. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν τον περιορισμένο χρόνο μας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρωτού ξεκινήσουμε έχω μία ανακοίνωση σε σχέση με τις ψηφοφορίες για το Money Market Fund. Έχουμε λάβει κάποια αιτήματα αναβολής της ψηφοφορίας λόγω της πολυπλοκότητας και της σημασίας της συμβιβαστικής πρότασης που είναι διαπραγμάτευση Ήρθα σε επαφή με τον εισηγητή. Προτείνω λοιπόν η ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 9 το πρωί. για τα money market funds, τα μηδέα κεφάλαια βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. Να καλωσορίσω τώρα τον Επίδροπο Τζόναθαν Χιλ, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι υπεύθυνο για την χρηματοοικονομική σταθερότητα, τι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίε και την Ένωση των Κεφαλαίων Ο κύριος Φεν Γκίκολτ. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα, Σα ευχαριστώ που μα δώσατε λίγο χρόνο για τα μηδά κεφάλαια των επενδύσεων. Ποιο είναι το πρόβλημα όμω, Παράλληλα με την ψηφοφορία διεξάγεται τριμερή διάλογος για την οδηγία περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Αν μπορούμε να συμβιβάσουμε τα δύο καλό είναι. Αλλά δεν μπορούμε να ψηφίζουμε ενώ ταυτόχρονα γίνεται ένα τριμερή διάλογο. Δεν μπορούμε να είμαστε και στα δύο μέρη ταυτόχρονα. Ναι, πράγματι. Θα προσπαθήσουμε να προγραμματίσουμε τον τριμερή διάλογο. Να καθυστερήσει λίγο ή να αναβληθεί ώστε να μπορούν να είναι όλοι εδώ. Όταν θα ψηφίζουμε για το MMF. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε εδώ τον Τζόναθαν Χίλ, επίτροπο Μοδιοκέ για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, που είναι και μία από τις ε, σημαντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής Juncker. Καλωσορίζουμε αυτή την ιδέα. Χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά κεφαλαίων επίσης, άρα αυτή η Ένωση κεφαλαγορών συμπληρώνει την πρωτοβουλία περί επενδυτικού προγράμματος, ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε χθε. Ο Επιτροπός μας παρουσίασε ένα πρώτο λιθαράκι, την πράσινη βίβλο. Είχαμε και έγγραφα διαβούλευσης ε. για το Prospectus Directive θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τη χάραξη του οδικού χάρτη θα έχουμε επικοδομητική συνεργασία. Σας δίνω μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων προς ε, τις ε, αντιδράσεις των πολιτικών ομάδων τη συνολική τους υποστήριξη στην πρόταση αυτή. Ήθελα όμως να έρθω και εγώ εδώ για να τα συζητήσουμε από κοντά, διότι πιστεύω ότι είναι καλύτερα πάντοτε να έχουμε μία μεσανταλλαγή απόψεων. Δεν έχω δυστυχώς πολύ χρόνο γιατί μεταβαίνω αμέσω μετά στι ΗΠΑ για να μιλήσω για τα θέματα τη διεθνού συνεργασία σε ζητήματα ρυθμίσεων. Ένα άλλο πολύ λεπτό θέμα που σα ενδιαφέρει με βέβαιο πολύ. Όπω είπε και ο κύριο Γκουαλτιέρη, αυτή είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία, ένα εμβληματικό έργο για αυτή την νέα αγορά κεφαλαίων στο πλαίσιο της όλης μας προσπάθειας για περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση. Αν τα 315 δισεκατομμύρια ευρώ αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα στόχο έχει να δώσει μια πρώτη όθηση για επενδύσει, η Ένωση των Κεφαλαιογόρων έχει ως στόχο να ενθαρρύνει επενδύσει μακροπρόθεσμε. Είναι ένα έργο, είναι ένα σχέδιο και για τα 28 κράτη-μέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι για κάποια νέα κράτη που δεν είναι τόσο αναπτυγμένες κεφαλαγορές του, ε, τα ωφέλη φαίνεται τα μεγαλύτερα και η δυνατότητα και το δυναμικό επίση πολύ μεγαλύτερο. Νομίζω βέβαια ότι η νέα αυτή η κεφαλαία αγορά στην Ευρώπη θα ε, ωφελήσει ολόκληρη την Ευρώπη, θα αναθερμάνει την οικονομία, θα στηρίξει επιχειρήσει, τι ευρωπαϊκέ και ιδίω τι μικρομεσαίε και τι νεοσυστήσει, οι νεοειδριόμενε εταιρείε. Θα είναι κάτι μεταξύ επενδύσεων, εθνικών ευκαιριών και επενδυτών. Θέλουμε το σύστημα για διαχείριση των κεφαλαίων να είναι πιο αποτελεσματικό. Σε πολλά μέρη τη Ευρώπη γνωρίζουμε ότι οι εταιρείε αγωνίζονται, παλεύουν να κτίσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται και τείνουν να βασίζονται κυρίως <clears throat> στις τράπεζες και όχι στις κεφάλαια αγορές ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου συμβαίνει το αντίθετο. Η... Το γεγονός αυτό ότι βασίζονται λύσεις στις τράπεζες καθιστά πιο ευάλωτη και την ευρωπαϊκή οικονομία όταν έχουμε ε, πιστοτική ασφυξία ή μείωση των δανείων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις. Και αυτό επηρεάζει και τη σταθερότητα βέβαια. Η Ένωση Κεφαλαγών θα είναι μια σημαντική αναβάθμιση σε ένα δίκτυο το οποίο διασυνδέει όσους χρειάζονται χρηματοδότηση με αυτούς οι οποίοι έχουν χρήματα να επενδύσουν. Βέβαια η Ευρώπη ήδη διαθέτει ένα αναπτυγμένο ε, χρηματοοικονομικό δίκτυο. Χρειάζεται όμως τώρα καλύτερες διασυνδέσεις ώστε αυτό το δίκτυο να γίνει ταχύτερο, να αναπτυχθεί περισσότερο και να είναι πιο αποτελεσματικό. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια κεφάλαιο αγορών η οποία στους ε, ελληνικού επενδυτέ θα δίνει πολλέ επιλογέ για το πού θα τοποθετήσουν τα χρήματά του. Θα δίνει επίση αξιοπιστία στην ακαιρότητα των αγορών για να προβούν σε αυτέ τι επιλογέ. Οι διαβουλεύσει ζητούν τι απόψει των διαφόρων φορέων για του καλύτερου τρόπου για να το πετύχουμε αυτό. Πώς ε, θα ε, επενδύουν είτε άμεσα είτε μέσω διαμεσολαβητών οι ελληνικοί επενδυτές. Και βέβαια και οι καταναλωτές θα πρέπει να αποκτήσουν εμπιστοσύνη. Η Ένωση Κεφαλαγορών ε, ουσιαστικά θέλει να συμπληρώσει το ρόλο των τραπεζών και όχι να τις αντικαταστήσει. Στόχος είναι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών λύσεων όχι η, η μίμηση αμερικανικών λύσεων. Φυσικά και ο κλάδος ε, θα ε, βοηθήσει πάρα πολύ, θα βοηθήσει τοπικές οικονομίες, τις τοπικές κοινωνίες. Είμαι βέβαιος ότι πολλές επιχειρήσεις βέβαια θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται μέσω τα δανείων. Θα υπάρξουν όμως άλλες επιχειρήσεις που σίγουρα ε, θα καλωσορίζουν περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης και σε χώρες που οι τράπεζες δεν δανείζουν βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις και οι δύο παλεύουν, αγωνίζονται. Άρα είναι καλό να υπάρχει αυτή η εναλλακτική χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, αν οι αγορέ επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη ήταν ανεπτυγμένε όσο οι αμερικανικέ επιχειρήσει θα μπορούσαν να αντλήσουν περαιτέρω 90 δι από το 2008 έως το 2013. Η δημιουργία μια σημεία αγοράς κεφαλαίων Σίγουρα είναι ένα μακρόπνο σχέδιο και φιλόδοξο σχέδιο ταυτόχρονα. Θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά. Κάποιες φορές ε, τα θέματα που θα μας απασχολήσουν ε, είναι πολύ ε, δύσκολα, φορολογική μεταχείριση, αφαιρεγγιότητα και πολλά άλλα. Άρα θα δούμε μεν πώ μπορούμε να προωθήσουμε τι επενδύσει και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά με το έγγραφο αυτό θα εξετάσουμε πιο προσεκτικά και κάποια από τα εμπόδια που πρέπει να εξαλείψουμε για να είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία των αγορών. Παραδείγματο χάρη τα εταιρικά ομόλογα που δεν έχουν οριστότητα και αυτό δημιουργεί προβλήματα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πολλέ φορέ προσπάθησαν να διευκολύνουν την κατάσταση. Θέλουμε να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα ε, τη περισσότερη τυποποίηση ε, είτε με ρυθμιστικέ παρεμβάσει είτε μέσω τραπεζικών δανείων. Επίση, περιβαλλοντική, κοινωνική, εταιρική διακυβέρνηση και τα σχετικά ομόλογα που συνδέονται με περιβαλλοντικά ζητήματα, κοινωνικά ζητήματα. Πάλι υπάρχει αυτή η τυποποίηση που καθοδηγείται από τις αγορές. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να στήριξουμε τη διαδικασία αυτή. Θέλουμε να δούμε επίσης πώς μπορεί να είναι πιο ελκυστικό και πιο εύκολο να επενδύουν και στις οσεκά οι διάφοροι επενδυτέ. Να δούμε τι γίνεται και με τα δυσυνεργά ταμεία. Και τι προβλήματα μπορούν να δημιουργούνται σε ορισμένε περιπτώσει. Σε περίπτωση απεργιότητα, τώρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορέ και σε ό,τι αφορά την ταχύτητα με την οποία λειτουργούν διάφορε νομικέ διαδικασίε. Και με του ε, συντελεστέ εσωτερικού. 450 δίσε θα μπορούσε να ανέλθει το ψηφαλές χρέος. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε για να μπορούν οι εταιρείε να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται από όλη την Ένωση. ή με μία ε να μπορούν να έχουν χρηματοδότηση πιο εύκολα, ή αποτεμιευτέ, οι καταθέτες να μπορούν επίσης να αποφελούνται από ένα ευρύ φάσμα προσιτών οικονομικά επενδυτικών δυνατοτήτων και για να προσελκύσουμε επενδυτές από όλες τις ε, χώρες του κόσμου να επενδύσουν στην Ένωση γιατί θα γνωρίζουν ότι είναι ασφαλείς οι αγορές μας, είναι σταθερές και αποτελεσματικές. Αυτό το, αυτή η πράσινη βίβλο λοιπόν σηματοδοτεί την έναρξη τριμερό, τρι, ε, συγγνώμη, τρίμηνων διαβουλεύσεων Περιμένω λοιπόν να ακούσω και από τους ευρωβουλευτές αλλά και από τους εθνικούς βουλευτές, κράτη-μέλη, ΜΜΕ, ΜΚΟ αλλά και από το χρηματοπιστωτικό τομέα και των 28 κρατών μελών τις απόψεις, διότι θα είναι ένα έργο, ένα σχέδιο και για τις 28 χώρες μέλη και θα πρέπει να φέρεις και τις 8 χώρες μέλη. Θέλουμε να ακούσουμε ποια είναι τα πρακτικά εμπόδια, ποια είναι η φραγμή, για να μπορέσουμε να τα επερπηδήσουμε ένα προς ένα. Βέβαια, είναι μεν μακροπρόθεσμο το όλο αυτό έργο, αλλά θέλω από νωρί να σημειώσουμε πρόοδο έξω και ξεκινήσανε δύο διαβουλεύσεις μαζί με την ε, Πράσινη Η μία αφορά την τυπλοποίηση και η δεύτερη αφορά την οδηγία προσπέκτου. Και θα σας πω τι ακριβώς κάνουμε. Με την πρώτη θέλουμε να δείξουμε μια ευρωπαϊκή αγορά υψηλής ποιότητας τυπλοποίηση που θα είναι διαφανής απλή και τυποποιημένη. Και αν μπορέσουμε αυτό να το πετύχουμε, μπορούμε να διευκολύνουμε τις τράπεζες να δανείζουν ε, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αν οι τετλοποίησεις των ΜΜΕ έχουν την ε, απόδοση έστω και του μισού που είχαν το 2007, αυτό θα μπορούσε να έρχεται σε 20 δις επιπλέον χρηματοδότηση. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε ε, στους παλιούς κακούς καιρούς ε, των στεγαστικών δανείων, αλλά θέλουμε να παρακολουθούμε την άκρος ε, πολύπλοκη διαδικασία και τα μέσα τιτλοποίησης. Πάντως διαβουλευόμαστε με το καλύτερο δυνατό τρόπο για να επιλέξουμε μια κατηγορία άκρος διαφανών απλών τυποποιημένων προϊόντων που θα συμβαδίζουν τις συστάσεις της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας θα ξεκινήσουμε αναθεώρηση και τη οδηγία προ επέκταση των ενημερωτικών δελτίων, δηλαδή ώστε και οι ΜΜΕ και άλλε επιχείρησει να μπορούν να ε, συλλέγουν πόρου σε κάθε χώρα. Θέλουμε να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο συγκεντρωσή κεφαλαίου, χωρίς να αφήσουμε σε κίνδυνο ε, τις επενδύσει. Τρεις μήνες θα διαρκέσουν διαβουλεύσει και ελπίζουμε να μπορέσουμε σύντομα να καταθέσουμε νομοθετικέ προτάσεις. Θα επανέλθω αργότερα φέτος με ένα σχέδιο δράση όπου θα αναφέρω τις προτεραιότητέ μας και τα επόμενά μας βήματα. Δεν υπάρχει μία απλή λύση ε, που θα ικανοποιεί τους πάντες. Θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή σε όλη την ε, θητεία αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Είναι μια καμπάνια, μια εκστρατεία που θα την ε, διαξαγάγουμε από κοινού. Περιμένω λοιπόν με ανυπομονησία τι ε, συνεισφορέ των μελών τη Επιτροπή σα και όχι μόνο σήμερα, αλλά και του επόμενου μέρε και τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Thank you, Commissioner. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Χιλ. Να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο για το πεντάλεπτο ερωταπαντήσεων στον πρώτο μιλητή, τον κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ, Επιτροπέ, για την σύντομη παρουσίαση τη πράσινη βίβλου από πλευρά τη ομάδα μα. Θέλω να σα πω ότι καλωσορίζουμε ιδιαίτερω την πρόταση αυτή και χαιρόμαστε για την ανταλλαγή απόψεων μαζί σα. Το ερώτημα που ανακύπτει για μα είναι το εξή. Όταν ξεκινάει τη δικασία πράσινη βίβλου και μα απεικονίσατε πώ οραματίζεστε τη μελλοντική διεκπαιρέωση, αναρωτιέμαι, έχουμε πραγματικά αυτό το χρόνο να περιμένουμε μέχρι τα τέλη της τρέχουσας θητείας, δηλαδή μέχρι ότου έχουμε νομοθεσία, γιατί τώρα διαπιστώνουμε ότι οι τράπεζες μειώνουν τους ισολογισμούς τους ε, λόγω και εξαιτία των πολλών προδιαγραφών που θέτουμε εμείς εδώ. Άρα βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία όπου χρειαζόμαστε κατεπηγόντως μια καλύτερα λειτουργούσα κεφαλαία αγορά. Και θα πρέπει να δράσουμε συγκεκριμένα, τώρα συγκεκριμένα. Έχω την εντύπωση ότι θέλετε να περάσετε αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να πουλήσει. Αναρωτιέμαι σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που θέλουν να κρατήσουν οι τράπεζες σε κάθε περίπτωση Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα της διάθεσης και πολύ κεφαλαίου κεφαλαίου σε αντιλοποίηση, σε ό,τι αφορά θέματα αντιλοποίησης, τι θα γίνει. Η απάντηση. Σε ό,τι αφορά τα θέματα νομοθεσίας, κατά πόσον έχουμε αρκετό χρόνο για να περιμένουμε. Δεν θέλω να περιμένουμε. Και καταλαβαίνω ιδιαίτερως ποια είναι, πόσο κατεπίγον είναι ο χαρακτήρας αυτής της εκστρατείας, δεδομένης δε της διαμόρφωσης των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εστίασης της θέσης ε, εργασίας και στην ανάπτυξη, κάθε μέρα αυτό που σκέφτομαι είναι τι μπορώ να κάνω στο δικό μου χαρτοφυλάκιο για να προωθήσω ακριβώς αυτή την προτεραιότητα των θέσεων επασχόληση και της ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την Ένωση Κεφαλαγορών τώρα η δική μου προσέγγιση δεν είναι. Ας κάτσουμε και θα συζητήσουμε πέντε χρόνια. Όχι. Η δική μου προσέγγιση είναι να ξεκινήσουμε καταρχάς με κάποια σωστή ανάλυση, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ποια είναι όλα τα εμπόδια και η δική μου προσέγγιση θα είναι να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε από, πάνω, από κάτω μέχρι πάνω την κεφαλαία αγορά. Ξέρουμε τους τομείς τιτλοποίησης και ξέρουμε πού μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Και εγώ πραγματικά ανυπομονώ να σημειωθεί πρόοδος. Και θέλω να ξεκινήσουν μαζί αυτές οι διαπραγματεύσεις με τις διαπραγματεύσεις και τις διαβουλεύσεις για την πράσινη βίβλο. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είσαστε ανυπόμονοι. Αλλά έχουμε μόλις ξεκινήσει ουσιαστικά και έχουμε δρομολογήσει πολλά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία τώρα, κατά πόσο θα υπάρξει νομοθεσία ή δεν θα υπάρχει νομοθεσία, νομίζω ότι σε κάποιους τομείς με πολύ σαφήνεια μπορώ να σας πω ότι χρειάζονται νομοθεσία. Αν ωστόσο βρούμε λύσεις που δεν προαπαιτούν νομοθεσία, όπως για παράδειγμα στους τομείς της ιδιωτικής επενδύσης, ε, των ιδιωτικών επενδύσεων, υπάρχει πρωτοβουλία από πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Αν λοιπόν υπάρχουν τέτοιες ε, λύσεις που μπορούν να σημειώσουν πρόοδο χωρίς νομοθεσία, είμαι ανοιχτός προς αυτές τις λύσεις, γιατί παίρνει πάντα χρόνο η νομοθεσία και θέλω εμείς ε, να προχωρήσουμε. Τώρα σε ό,τι αφορά την τυπλοποίηση, Ελπίζω ότι όλοι όσοι έχουν διαφορετικέ απόψει σε ό,τι αφορά την τυπλοποίηση είναι πιο επεκτικοί ή πιο θετικοί να μας δώσουν τις απόψεις τους, γιατί θεωρώ ότι αν περάσει σωστά το σύστημα αυτό, μπορούν να βοηθηθούν οι τράπεζες προκειμένου να δανείσουν πιο πολύ στην οικονομία. Αυτό φυσικά θα είναι επωφελές και τις ε, τράπεζες, για τις τράπεζες αλλά και επικριτές για τις επιχειρήσεις που θέλουν τις επενδύσεις. Ευχαριστώ. Η Νίνα Τζιλ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε Χίλ για την παρουσίασή σας. Καλωσορίζω την επισήμανση ότι πρέπει να ε, διαθετήσουμε την αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναφέρατε μια σειρά από ζητήματα που ήθελα και εγώ να θίξω, όπως την τιτλοποίηση. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν το στόχο επίτευξης συνολικής και ομαδικής προσέγγισης στην διπλοποίηση. Όμως δεν επισημαίνει πώς θα υπάρχει στις δευτερογενείς αγορές ρευστότητα σε βάθος για να υπάρχει ε, σαφήνεια και για την έκδοση και για τις επενδύσεις. Λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα και για τους 28. Όμως Ρεαλιστικά, πώς πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει διαφορά στην πράξη για μια μικρομεσαία επιχειρήση λόγω χάρη στην Πορτογαλία και μια άλλη στη Γερμανία ή στην Ελλάδα. Οι ανάγκες τους είναι πολύ διαφορετικές. Οπότε σημαντικό είναι να αλλάξουμε λιγάκι το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Πρέπει πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Δηλαδή, συνήθω πάει κανεί στην τράπεζα για να ζητήσει χρήματα. Είναι τόσο απλό. Και έπειτα, μια πραγματική πρόκληση θα είναι πώ να ξεπεράσουμε το θέμα των ε, αλληλένδετων συμπερόντων. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για το θέμα των χρηματαγορών. Και βλέπω ότι αυτά τα αλληλένδετα συμφέροντα τα, ε, των είναι πάρα πολύ ισχυρά στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν την προτινόμενη νομοθεσία από το να γίνει πραγματικά νομοθέτημα. Πώς μπορούμε λοιπόν τη διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, να την προστατεύσουμε από τον ε, ενδιαφερόμενο αυτό κλάδο και να είναι αδιάβλητη διαδικασία, όπως είπε και ο κύριος Φέρμπερ. Πώς μπορούμε να δράσουμε με ταχύτητα σε αυτές τις προτάσεις. Συμφωνώ κατά πολύ με την ουσία των παρατηρήσεών σας. Δηλαδή, δεδομένου ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει σε διαφορετικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαφορές και να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Θα υπάρξει μια σειρά από μέτρα που πρέπει να αναλάβουμε. Και αν είναι τα σωστά, συνδυασμένα θα ε, διευκολύνουν. Ένα μέρο τη απάντηση είναι πώς μπορέσουν οι επενδυτές να λαμβάνουν εύληπτες πληροφορίες για μια μικρομεσαία στην οποία μπορεί να θέλουν να επενδύσουν. Προς στιγμή, με τις αποκλίνουσες πληροφορίες θα μπορούσε κανείς να ρωτηθεί γιατί ένας επενδυτής στη Γαλλία να βρει νόημα στο να επενδύσει σε μια εταιρεία high-tech στις χώρες της Βαλτικής. Το θέμα είναι λοιπόν να έχουμε τυποποιημένε πληροφορίε ώστε να μπορεί ο επενδυτή να εντοπίσει τον κίνδυνο. Κάποιες βεβαίως είναι θέμα νοοτροπία. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τα πάντα για και να πει ότι μπορεί κανείς να περάσει από την πλήρη απουσία επιχειρηματική νοοτροπία στην απόκτησή τη. Θα χρειαστεί χρόνο. Κάποιοι Χρειάζεται να επικεντρωθούν στη χρηματοδότηση, αλλά η βασική μου παρατήρηση είναι ότι πραγματικά ευνηδιάστηκα συζητήσει που είχαμε μια σειρά από εκπροσώπου μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μια σειρά από εκπροσώπου κρατών μελών. Αυτοί που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένε αγορέ κεφαλαίων και πιο ομοιογενές ε, τοπίο και σκηνικό προς τις εταιρείε είναι οι πλέον ενθουσιώδης για τις ε, δυνατότητες που τους προσφέρει η αγορά κεφαλαίων. Ε, γι' αυτό λοιπόν τονίζω ότι αυτό το εγχείρημα αφορά και τους 28. Ως προς τις ειδικότερε ερωτήσεις για την τυπλοποίηση, προφανώς είναι εύστοχες, γι' αυτό και έχουμε διαβολεύσει σχετικά, πρέπει να έχουμε μια λογική και σταθερή προσέγγιση για να ορίσουμε το σωστό πλαίσιο. Και έτσι πρέπει τα συμφέροντα αυτά να τα δούμε, τα συμφέροντα της διαπλοκής. Πρέπει να τα δούμε από διαφορετικές σκοπιές. Είναι εμπορικά, είναι χρηματοοικονομικά, και πολλοί σε όλη αυτή την αλυσίδα έχουν και εθνικά συμφέροντα. Μιλάμε για κράτη σε κάποιε περιπτώσει. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνει κανεί, και εγώ θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια σχετικά, είναι να εντοπίσει το πρόβλημα, να προτείνει λύσει και μετά να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Δηλαδή, με τα κατάλληλα επιχειρήματα να προσπαθήσει να υπερβεί τα εμπόδια να ακούσει αυτό που έχουν να πούν οι ενδιαφερόμενοι, αλλά να διαμορφώσει την πλέον ευσταθούσα άποψη για το τι οφείλει να πράξει. Αυτή θα είναι και η προσέγγιση μου. Thank Σας ευχαριστούμε. Τώρα για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Ρούμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Χιλ. Υπάρχουν πολλά προγράμματα για την πράσινη βιβλίο τη ε, Ένωση Αγορά Κεφαλαίων και το στηρίζουμε από την δική μα ομάδα με έμφαση στο ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα για τι επιχειρήσει που μπορούν να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Οι Financial Times σα ανέφεραν σαν υδραυλικό με μια παρομοίωση, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα παραπλανητικά τεχνικά ερωτήματα στην Τραπεζική Ένωση και την αγορά κεφαλαίων. Βλέπω ότι έχετε τρεις προτεραιότητες. Την οδηγία για τα ενημερωτικά δελτία, την οδηγία για τη διαφάνεια, πρέπει να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθο και εγώ ήθελα να ρωτήσω τα εξή. Ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο στο θέμα των μικρομεσαίων πρώτων. Το θέμα είναι πώς να φτάσουν τα χρήματα στις μικρομεσαίες, αλλά θα επικεντρωθούμε μόνο στι καινοτόμε ε, και γοργά αναπτυσσόμενε μικρομεσαίες, αυτές που δρούν πολύ σε εθνικό επίπεδο ή και στις παραδοσιακότερες, αυτές που είναι ο ιστό της οικονομίας μας, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη είναι αν έχετε την πρόθεση να αναλάβετε δράση ώστε βασικά τμήματα τη νομοθεσία για την αγορά κεφαλαίων όπω η MIFID και η SSDR, ο κανονισμός SSDR, μπορούν να διαρθρωθούν μεταξύ του, ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων τη Ένωση και να υπάρχει περισσότερη ρευστότητα σε αυτή την αγορά για τις ε, επιχειρήσει όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και ευχαριστώ για τη στήριξή σα. Ευχαριστώ που μου θυμίζετε ότι είναι σαν να μην ε, για την Ένωση Αγορά Κεφαλαίων. Η σύζυγός με ξεπλάγει όταν ε, ε, με περιέγραψε ένα συντραυλικό γιατί γενικώ δεν είμαι πολύ ταλαντούχο στα δωρέματα στο σπίτι. Θεώρησε λοιπόν ότι είναι πολύ ειρωνικό το σχόλιο. όσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσει, νομίζω ότι θέσατε πολύ σωστά την πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι διαφορετικέ επιχειρήσει σε διάφορα στάδια ανάπτυξη, από τι νεοδριούμενε μέχρι τι μεγάλε επιχειρήσει, είναι περιπτώσει που θέλουμε να έχουν τις ροές ε, χρηματοδότησης που τους πρέπουν. Προ στιγμήν Υπάρχουν πολύ καλέ επιχειρηματικέ ιδέε που επιτρέπουν να φτάσει η επιχείρηση σε ένα συγκεκριμένο μέγεθο, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί κι άλλο συχνά. Οπότε χρειάζεται στήριξη από τράπεζα ή από την αγορά κεφαλαίων. Πολλέ φορέ πάνε ε, στι ΗΠΑ για τι τοποθετήσει του ή για το κεφάλαιο κινδύνου. Ε, τι αξιοποιούν οι ΗΠΑ λοιπόν. Αυτέ τι ε, αρπάζουν και όχι εμεί. Με, με τα προλικά έσοδα και τι θέσει απασχόληση που θέλουμε να δημιουργήσουμε και χάνουμε. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτή την βιώσιμη ανάπτυξη που θέλουμε να δημιουργήσουμε και τις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης που χρειαζόμαστε. Πολλές φορές υπάρχουν οι, τα ιδιωτικά αξιόγραφα, τα κεφάλαια κινδύνου και οι επενδυτές κινδύνου. Όλα αυτά ανθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπάρχει ένα δυναμικό ανάπτυξης που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Όμω για την παρατήρησή σα για την υπάρχουσα νομοθεσία και πώ διασφαλίζουμε ότι εν γέννη η νομοθεσία μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη. Νομίζω αυτό είναι ευθύνη όλων μας, από κοινού. Νομίζω το επίτευγμα της τελευταίας πενταετίας με την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτική και τραπεζικής κρίσης και την ε, νομοθετική ε, οικοδόμηση και αναδιάρθρωση που κάναμε ήταν εντυπωσιακή, με πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως νομίζω ότι είναι θέμα κοινή λογική να πάρουμε λίγη απόσταση από όλο αυτό και να δούμε αν όλε οι πτυχέ, οι παράμετροι αυτή τη αναδιάρθρωση ήταν ε, οι κατάλληλε. Το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζω τώρα είναι η έλλειψη ανάπτυξη και θέσεων απασχόληση. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το θέμα είναι λοιπόν αν έχουμε βρει το σωστό σημείο ισορροπία. Εκεί θα πρέπει να, από αυτή την άποψη θα πρέπει να αντικρίσουμε το όλο θέμα. Και με, το, με την οδηγία Solvency 2 και την κάλυψη ρευστότητας, θα πρέπει να χαλαρώσουμε, όπω είδαμε, τι απαιτήσει μα κάπω και τι υποχρεώσει που επιβάλλουμε με έναν τρόπο λίγο πιο φιλικό προ την ανάπτυξη. Από αυτού θα επανέλθω. Σα ευχαριστώ. Η Σιλβή Γκουλάρα από την Άλντα. Καλημέρα σας, Επίτροπε. Ευχαριστώ που ξανάρχεστε εδώ και ευχαριστούμε για τη δουλειά σα, που είναι μια πολύ καλή βάση. Η ομάδα μα χαιρετίζει την πρωτοβουλία σα. Τρει πολύ σύντομε παρατηρήσει. Πρώτον, τα αναφέρατε ήδη το χρονοδιάγραμμα ε, επιτεχμένο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση μεταξύ της γενικής σας αιτιολόγησης, jobs and growth, και του χρονοδιαγράμματος που έχετε προβλέψει. Όλα, ε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα είναι πολύ σημαντικό. Έχετε αναλάβει καθήκοντα βέβαια, αλλά το πρόγραμμα εργασιών ε, φτάνει, ανάγεται στο 1999 όπως θα λέγαμε στο Βέλγιο με την βελγική αναφορά του αριθμού. Ε, εδώ λοιπόν πώς θα προωθήσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εδώ υπάρχει ένα S παραπάνω νομίζω στις προτάσεις σας. Capital Markets Union, δηλαδή πολλές αγορές κεφαλαίων της Ένωσης ή μία ένωση, μια ενιαίας αγοράς κεφαλαίων. Νομίζω, αν ο στόχος σας είναι να πάρετε κάποια μέτρα που θα επιτρέψουν οι αγορές να παραμείνουν απομονωμένες μεταξύ τους, θα χάσουμε την ευκαιρία να έχουμε πραγματική χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν τι προτείνετε για να υπερβούμε τα εμπόδια ε, αυτοχαρακτηριστήκατε ως υδραυλικός. Εγώ δεν έχω δει πολλούς υδραυλικούς να προτείνουν ενώσεις, ασχολούνται με τις διασωληνώσεις περισσότερο. Εδώ λοιπόν ε, έχουμε μια διάσταση πανευρωπαϊκή Θεωρείτε ότι η ΕΣΜΑ πρέπει να έχει εδώ έναν ενισχυμένο ρόλο. Ε, μπορούμε να καταργήσουμε κάποιου εθνικού φραγμού όπω έγινε με την Τραπεζική Ένωση. Διότι βλέπουμε τι παραλληλισμό μπορεί να κάνει κανεί. Με την Τραπεζική Ένωση, ε, στην Ευρωζώνη τουλάχιστον, φτάσαμε μια μεγάλη, ένα σημαντικό επίπεδο ενοποίηση. Και μια τελευταία παρατήρηση. Το αναφέρει και το έγγραφό σα, αλλά είναι και το θέμα τη νοοτροπία στην Ευρωζώνη προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι που ακούγονταν πολύ ωραίο στα χαρτιά. Πολύ ορθολογιστικό, πολύ λογική πρόταση ακούγεται το ευρώ. Στα χαρτιά είναι τέλεια. Όμω, όταν έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα με πολίτε που δεν έχουν την ίδια αντίληψη για το τι είναι ένα νόμισμα, ποια είναι η ανεξαρτησία μια κεντρική τράπεζα και η σχέση του με την οικονομία διαφέρει, θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Ότι είναι ιδιωτικό τομέα θεωρείται ύποπτο από ένα μέρο τη κοινή γνώμη, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν τη συνήθεια να πηγαίνουν στι αγορέ κεφαλαίων. Φοβάμαι λοιπόν χωρίς να έχω καμία κακή προαίρεση, ότι μπορεί να σκοντάψουμε στο θέμα των πολιτιστικών διαφορών. Ναι, να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση και καταλαβαίνω τι λέτε για την πολιτισμό και καταλαβαίνω επίσης και δεν είμαι αφελής. Δεν πιστεύω ότι μία νομοθεσία ή οποιαδήποτε άλλο μέτρο ξαφνικά θα αλλάξουν τη συμπεριφορά εκατομμυρίων ανθρώπων και θα αλλάξουν οτροπίες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία εκατοντάδες χρόνια. Κοιτώντα τι ευρωπαϊκέ κεφαλαίε αγορέ, ε, διαπιστώνω ότι υπάρξει, υπάρχει ανάπτυξη. Ή έχει υπάρξει ανάπτυξη και νομίζω ότι υπάρχει και άλλη όρεξη, άλλη ορμή και πρέπει να, την, να επαφαληθούμε από αυτήν. Να βρούμε τα στοιχεία που μας εμποδίζουν και την εμποδίζουν από το να αναπτυχθεί πιο γρήγορα. Γι' αυτό που αναφέρατε για την ταχύτητα τώρα. Εγώ θα πάω ακόμα πιο πίσω από το 99, στη συνθήκη της Ρώμης που όρισε την ε, φιλοδοξία της ενιαίας αγοράς, της ενιαίας κεφαλαγοράς. Πάνω από μισό αιώνα λοιπόν μας απασχολεί το θέμα αυτό. Συμπεραίνω δε διάφορα πράγματα. Καταρχάς, ότι δεν θα πρέπει να είμαι αλαζονικός, να μην επιδείξουμε ύβρι για το τι μπορούμε να πετύχουμε. Δεύτερον, πιστεύω, πιστεύω στις πολιτικές, στην πολιτική. Όταν αλλάζουν οι συνθήκες και παρουσιάζονται μια ευκαιρία και υπάρχει και το κατάλληλος ε, αυταρισμός, ε, θα πρέπει να αντράτουμε τις ευκαιρίες, γιατί τότε έχουμε την ευκαιρία να σημειώσουμε πρόοδο για να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε μια κοινή αγορά. Αγορά, όχι αγορές για τα κεφάλαια. Στο θέμα που αναφέρεται σε σχέση με τη φιλοδοξία και την ταχύτητα, συμφωνώ απόλυτα. Ελπίζω όλοι μας δε να έχουμε υπόψη μας ανά πάσα στιγμή τι σημασία έχει η ταχύτητα προκειμένου να προωθούμε τα στοιχεία αυτά. Η άποψή μου όμως για κάποια στοιχεία με οδήγησε την ανάπτυξη της φιλοδοξίας, γιατί πιστεύω ότι αν σημειώσουμε μία πρώτη πρόοδο, μπορούμε να δώσουμε μία ορμή, να διαμορφώσουμε μία γενική κατεύθυνση και κατά συνέπεια να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια σε αυτό που συγκεκριμένα αναφέρατε τώρα για την ΕΣΜΑ για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει δράση εκεί. Στην πράσινη βίβλο τίθεται το θέμα της εποπτείας, κατά πόσον χρειάζεται να υπάρχει καλύτερη σύγκληση, κατά πόσον πρέπει να υπάρχει πιο πολύ σύγκληση μεταξύ των διαφορών αρχών ή κατά πόσον υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Να ταξιδάσουμε τα ερωτήματα αυτά. Δεν έχω δει κάποια αντιτράταχτα τεκμήρια που να καταδεικνύουν ότι οι θεσμικοί οι θεσμικοί ρυθμίσεις που έχουμε προσφάτως αποφασίσει θα πρέπει να αλλάξουν, να προσαρμοστούν, αλλά να το εξετάσουμε στα πλαίσια της πράσινης βίβλου. Έχετε αυτή το ερώτημα άλλωστε. Και να δούμε προς ποια κατεύθυνση μας οδηγούν τα δεκμήρια. Ευχαριστώ. Ο Φάμπιο Ντεμάζη από την ΚΟΕ. Ναι, όπως είπε και ο Μαρκός Φέρμπερ και σε Βίγκουλαρ ε, για θέματα της Ένωσης Κεφαλαγορών, εγώ θα σας ρωτήσω για κάτι άλλο και θα συμφωνήσει και η γυναίκα σας που έχει εμπειρία σε ό,τι αφορά το έργο των υδραυλικών στα σπίτια. Εγώ ήθελα να κάνω δύο γενικά σχόλια για την Ένωση Κεφαλαγορών. Καταρχάς, πιστεύω ότι τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε στην παρούσα φάση στην Ευρώπη δεν αποτελούν πρόβλημα ρευστότητα. Έχουμε πολλή ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, αλλά οι πιστώσεις δεν ε, κυκλοφορούν επαρκώς και κάθε τραπεζίτη θα σας πει ότι ε, οι πιστώσεις δίνονται όταν υπάρχει και σωστή ζήτηση. Υπάρχει θέμα ζήτηση, λοιπόν. Δεν έχουμε πρόβλημα ρευστότητας, έχουμε πρόβλημα ζήτησης για επενδύσεις. Και το πρόβλημα δεν είναι σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κ. Βαρουφάκης και αυτά που είπε ο κ. Σόιμπλε, τι είναι να συμφωνήσω να μην ε, συγκρίνουμε επίσης ε, τις ε, κεφαλαγορές των ΗΠΑ με αυτές της Ευρώπης. Μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα, γιατί είναι πολύ διαφορετική η παράδοση. Εμείς βασιζόμαστε πολύ πιο πολύ στην παραδοσιακή πίστοση προς τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό το γεγονός. Τρίτον, να πω ότι υπήρχαν κάποια στοιχεία στην πρωτοβουλία με τα οποία συμφωνώ, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ε, οδηγία για τους προσπέκτορς και την ανάπτυξη των ε, αγορών ιδιωτικών τοποθετήσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι οι πραγματικές οικονομίες θα πρέπει να κοιτάξουν το θέμα της αντικυκλικής ε, κίνησης. Δεν είμαι φυσικά κατά της ε, απλής και διαφανούς δυσλοποίησης, ε, αλλά το θέμα του της ε, εξέτασης σε επίπεδα, σε μερίδες, δεν ξέρω πώς μπορώ να αντιδράσω σε αυτό. Και τέλος, να πω το εξής, ότι από ό,τι ακούσαμε από τους εμπλεκούμενους φορείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν φυσικά πολλούς θεωρούν ότι η διπλοποίηση είναι κάτι πολύ ακριβό, πολύ δύσκολο. Πείτε μου ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν από αυτού. Καταρχάς πιστεύω ότι σωστά τα λέτε. Υπάρχει η πλευρά της ζήτησης και η πλευρά της προσφοράς. Εγώ εστιάζομαι στον τομέα της προσφοράς στη δουλειά μου και πιστεύω ότι και τα δύο θα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Αυτό σκοπεύω να κάνω. Πολύ συμφωνώ με αυτό που είπατε. Ότι δεν θα πρέπει σκοπός μας να είναι να πιστέψουμε ότι πρέπει να εισαγάγουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το αμερικανικό στην προκειμένη περίπτωση. Πολύ σωστά επισημάνατε ότι έχουμε διαφορετική ιστορία, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικούς νόμους, διαφορετικά εργαλεία. Και συμφωνώ απόλυτα. Αν υπάρχουν χρήσιμα παραδείγματα από τα οποία μπορούμε να επωφεληθούμε, ασφαλώς να το πράξουμε αυτό. Τα παραδείγματα που έχω χρησιμοποιήσει έως τώρα για, το διάφορα, διαφορετικά μεγέθη, αν θέλετε, των αγορών μας, είναι ενδεικτικά για να καταδείξω ποια θα ήταν ενδεχόμενα ωφέλη, αν πετύχουμε. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια μακρά και επιτυχή παράδοση στο τραπεζικό μας σύστημα και σε καμία περίπτωση δεν προτίθεμαι να αντικαταστήσω την μακρά αυτή παράδοση. Όχι. Προσπαθώ να τα συμπληρώσω. Και νομίζω ότι σε κάποια τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα πράγματα πηγαίνουν καλά, ο κόσμο θέλει να συνεχίσει την καλή συνεργασία με τι μικρέ τράπεζε. Αλλά σε άλλα τμήματα όπου δεν υπάρχει σωστή λειτουργία, να βρούμε εναλλακτικέ μορφέ χρηματοδότηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστή αυτή η κατεύθυνση. Η τυπλοποίηση, όσο είναι διαφανής και απλή, συμφωνώ μαζί σας. Αν έχετε την αίσθηση ότι πρέπει να το εξετάσουμε, εντάξει, για το τώρα πώς θα κινηθούμε συγκεκριμένα, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα συγκεκριμένα, θα πρέπει να τα βρούμε αυτά στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές γνωμοδοτήσεις που υπάρχουν από πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της ε, Αγγλίας και το Όσλο, η Βασιλεία. Τα εξετάζουν όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ισόρροπη η προσέγγιση μας και να κοιτάξουμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε ένα σωστό πλαίσιο το οποίο θα απαλύνει και θα καθησυχάσει τις ανησυχίες σας και θα επιτρέψει παράλληλα στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν την τυπλοποίηση προκειμένου να διευκολυνθούν στην παροχή πιστώσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που το επιθυμούν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Σβέν Γκίγκολτ από τους Πράσινους τώρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι με πολύ ενδιαφέρον άκουσα αυτά που είπατε για τα μαστορέματα, γιατί όταν σας πρωτοσυνάντησα μου είπατε ότι ασχολείστε με την Κυπουρική. Τώρα ε, προσπαθείτε να συμφιλιώσετε την Κυπουρική χωρίς να ασχοληθεί το ίδιο, ε, χωρίς να ε, λερώσετε τα χέρια σας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί και εγώ δυσκολεύομαι να τα πετύχω αυτά τα δύο. Σε ό,τι αφορά την Ένωση Κεφαλαίου και ε, εν γέννη είναι μια καλοδεχούμενη πρωτοβουλία για την ομάδα μας, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη. Επίσης, ε, πολλές από τις ιδέες ε, της Πράσινη Βίβλου τις επικροτούμε. Συγκεκριμένα θα σας ενθαρρύναμε να παραμείνετε αποφασιστικός και σταθερός σε ό,τι αφορά απλά λιανικά προϊόντα. Ακούμε ότι υπάρχει ήδη έντονη αντίσταση και αυτό είναι πολύ κατανοητό. Αν έχουμε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία θα είναι απλά και ε, ρυθμισμένα. Θα είναι καλύτερες οι συμφωνίες για τους ε, καταναλωτές. Εμείς θέλουμε να σας ζητήσουμε να παραμείνετε αποφασιστικός ως προς αυτό το σημείο. Κρίμα βέβαια είναι κάπως ότι σε επίπεδο αρχών θα μπορούσε το να είναι πιο ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συμφιλειώσουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαίου Αγορών με τις ευρωπαϊκές αξίες. Τι εννοώ με αυτό ο προσανατολισμός σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και ο προσανατολισμός προς ε, αηφορία, δηλαδή κοινωνικά περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε λεγόμενα ίσως προϊόντα όπως τα green bonds, τα πράσινα ομόλογα, αλλά η κεφαλαία αγορά συνολικά θα πρέπει να υπηρετεί τις ευρωπαϊκές αξίες και να μην αναζητεί ε, το βραχυπρόθεσμο κέρδος για τους μετόχους. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα συμπεριλάβουμε στις πρωτοβουλίες μας και να μην ε, παράγουμε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τι ένα τελευταίο ερώτημα. Συμφωνώ μαζί σα ότι οι εταιρείε χρειάζονται διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης, περισσότερες πηγές χρηματοδότησης. Με τη ρυθμιστική επίθεση, αν θέλετε, είδαμε ότι οι μικρές τράπεζες που μπορεί να τα πηγαίνουν καλά σε κάποιες ε, χώρες Ευρώπης αντιμετωπίζουν πλέον περισσότερες δυσκολίες. Θα ήσασταν ανοιχτό στην ανάπτυξη παράλληλα με την ε, Ένωση Κεφαλαιογόρων μιας πρωτοβουλίας που θα στηρίζει τις μικρότερες τράπεζες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το βάρος και να αναπτύσσουν ε, τραπεζικές υπηρεσίες που δεν θα έρχονται σε αντίφαση με την ε, Ένωση Κεφάλαιο θα είναι πιο πολύ κοινωνικές υπηρεσίες. Ο Επίτροπος, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ υδραυλικού και κυπουρού. Ε, η κυπουρική είναι εύκολη δουλειά. Ε, σκάβεις μόνο. Δύσκολα μπορεί να κάνεις μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Πολύ περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει αν τα κάνεις ε, στραβά. Ε, ο παρός και πουρός. Τώρα, λιανικός επενδυτής. Είναι σημαντικό να τον έχουμε υπόψη μας και κάτι άλλο το οποίο είναι εκτός ίσως ε, των κεφάλαιων αγορών, αλλά θα ήθελα να εργαστώ πάνω σε αυτό και θα ήθελα την υποστήριξή σας, είναι το να δούμε γενικά τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το κατά πόσον μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα τις αντιμετωπίσουμε υπό το πρίσμα του πώς μπορούμε να έχουμε αύξηση ανταγωνισμού, φθηνότερε τιμές, καλύτερα προϊόντα από τους καταναλωτές. Να το βλέπουμε από την άλλη πλευρά του τηλεσκοπίου και όχι από πάνω προς τα κάτω, από τη στρατόσφαιρα προς τα κάτω, αν θέλετε. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω λοιπόν εκτός αυτής της παρουσίας της και θα σας αναφέρω τον προβληματισμό μου και τις προτάσεις μου αργότερα, στη διάρκεια του έτους. Ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, η φορεία, το μακροπρόθεσμο επίπεδο, συμφωνώ. Και νομίζω ότι είναι και ένας από τους τρόπους με τον οποίο μπορούν οι κεφαλαιογορές να βοηθήσουν. Αν δηλαδή έχουμε επενδύσει από μακροχρόνιου επενδυτέ όπω είναι ασφαλιστικέ εταιρείε, τα εξωτερικά ταμεία, και διαθέσουμε τα κονδύλια σε έργα υποδομών, μακροπρόθεσμε επενδύσει. δηλαδή. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για να πετύχουμε την αηφορία για την οποία μιλήσατε. Υπάρχουν βέβαια και πιο συγκεκριμένα προϊόντα. Πράσινα ομόλογα είπατε, τέλο πάντων να μην πούμε προϊόντα, όπω θέλετε πείτε το. για κάποιες επιχειρήσεις αυτό έχει νόημα και από εμπορικής πλευράς και από κοινωνικής και περιβαλλοντικής. Για τις τράπεζες και τις μικρότερες τράπεζες νομίζω ότι κάποια κράτη-μέλη εξετάζουν αυτό το τομέα που αναφέρατε και με τα χαράς να συνομιλήσουμε και να το δούμε και από την πλευρά των τραπεζών. Είναι λίγο εκτός βέβαια της, ε, του πεδίου της Ένωσης Κεφαλαίου, αλλά γιατί να μην την ε, προωθήσουμε την ιδέα αυτή, να τη διερευνήσω ευχαρίστω, γιατί η βασική μου προσέγγιση πάντοτε είναι πώς μπορούμε πρώτον να εξισορροπήσουμε την ενθάρρυνση ε, της ανάπτυξης με τη μετρίαση των κινδύνων. Εγώ δεν πιστεύω στο ότι ένα μέγεθος είναι καλό για όλους, πρέπει να είναι διαφοροποιημένο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την ευθυντή Μάργο Πάρκερ. Uh, Καλημέρα σας, Λόρδε Χιλ. Να μην σας θυμίσω ότι ο Γιούνκερ και ο Κατάινεν είναι τα σας. Εάν, όπως λέτε, δεν έχει τίποτε ιδιαίτερο το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό ποιε συνθήκες φαντάζεστε ένας Βρετανός Πρωθυπουργός να εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και επιπλέον να πω το εξή. Δεδομένων των ευθυνών σα για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη χρηματοοικονομική μάλλον σταθερότητα, φαίνεται να, να, να ανακουφιστήκατε την περασμένη εβδομάδα όταν το πρόγραμμα της Ελλάδας προτάθηκε. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τι απόψει σα. Uh, ε, well, I, on, on... Κοιτάξτε, για την πρώτη σα ερώτηση δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο το Ηνωμένο Βασίλειο η Βρετανία. Όμως η δική μου παρατήρηση για την αγορά, για την Ένωση της Αγοράς Κεφαλαίων στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που το στηρίζω θερμά, είναι ότι η Ένωση Αγοράς Κεφαλαίων θα πρέπει να ισχύει και για τα 28 κάτι μέλη και έπειτα πολλοί μου είπαν και με ρώτησαν αν είναι αυτό ένα εγχείρημα που αφορά και το City του Λονδίνου. Η απάντησή μου είναι ότι εάν λειτουργεί εύρυθμα η αγορά είναι ανοιχτή, εάν οι επιχειρήσεις είναι ισχυρές και προσφέρουν καλές ανταγωνιστικές υπηρεσίες, θα έχουν ευκαιρίες. Αυτό θα ισχύει για όποιο σημείο της Ένωσης και αν είναι η έδρα τους. Σε ό,τι αφορά τις γενικότερες παρατηρήσεις σας για την κατάσταση στην Ελλάδα και ούτω καθεξής, Νομίζω η σύντομη τοποθετησή μου είναι αυτή. Όντως, τα μέλη του Eurogroup εν γέννη και η Ελλάδα συγκεκριμένα είναι αποφασισμένοι να βρουν έναν τρόπο συμβιβασμού μεταξύ των διαφόρων διαφωνιών που υπάρχουν και να καταλήξουν σε μια λύση που θα τους επιτρέψει να τιμήσουν να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του και να επιτρέψει στην Ελλάδα να παραμείνει μέλο τη Ευρωζώνη. Αυτό είναι και μια σαφή επιθυμία και τη Ελλάδα, αλλά και του υπόλοιπου τη Ευρωζώνη. Θέλουμε να παραμείνουν μαζί μα. Ευχαριστούμε η Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ για τις παρουσιάσεις σας και για τα θέματα κεφαλαίων αγορών. Είπατε ότι επί 50 χρόνια μας απασχολεί το θέμα αυτό από τη συνθήκη της Ρώμης. Σίγουρα όμως σήμερα είναι πολύ επικριτό θέμα αυτό ιδιαίτερα από το ξέσπασμα της κρίσης επειδή η Ευρώπη αντιμετωπίζει 400 δισεκατομμύρια έλλειμμα επενδύσεων. Και σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να αφαιρθώ στην ερώτησή μου σε ό,τι αφορά την μακροπρόθεσμη επένδυση των θεσμικών επενδυτών. Στην πράσινη βίβλο αναφέρεται ότι έχουμε 12.000 δισεκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά ε, συντάξει που διατίθενται στου θεσμικού επενδυτέ, τα οποία μπορούν να εισρέψουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ευρώπη έχει 350 δισεκατομμύρια προβλέψει με το σχέδιο Juncker, το οποίο όμω είναι ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο, δεν έχει μακροπρόθεσμε ε, βλέψει. Ερωτώ λοιπόν προ ε, τη δική σα κατεύθυνση. Ένα από του στόχου που αναφέρατε στο σχέδιο είναι και ή δημιουργία μακροπρόθεσμων επενδυτικών ταμείων. Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε ποια κίνητρα θα δημιουργήσετε προκειμένου οι θεσμικοί επενδυτές, ιδιαίτερα τα συνταξιδοτικά ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, να διοχετεύσουν τα χρήματα αυτά στα ευρωπαϊκά έργα και κατά δεύτερον, πώς θα προσεγγίσετε τον στόχο των ευρωπαϊκών μακροπρόθεσμων επενδυτικών ταμείων προκειμένου να δημιουργηθούν και να προωθήσουν ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Well, uh, Νομίζω ότι στο ερώτημα του πώς θα ενθαρρύνουμε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ε, αυτό ασφαλώς αποτελεί ένα κεντρικό ζήτημα στους τομέες που εξετάζουμε σε ό,τι αφορά τα θέματα κεφαλαγορών και ένωσης κεφαλαγορών. Προσφάτως λοιπόν ε, στα τέλη της περιορισμένης χρονιάς ε, λάβαμε μέτρα για τα ευρωπαϊκά επενδυτικά ταμεία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς αυτά θα αρχίσουν να λειτουργούν σωστά. Θεωρώ όμως ότι αν μπορέσουμε να κάνουμε την Ένωση Αγορών να λειτουργεί καλύτερα, οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις που μπορούν να κάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα συνταξιβατικά ταμεία, σε μακροπρόθεσμα έργα, όπως τα έργα υποδομών, όπου υπάρχει ανάγκη να υπάρχει κάποια μακροπρόθεσμη σιγουριά των αποτελεσμάτων, των αποδόσεων. Αν λειτουργήσουν λοιπόν αυτά καλύτερα, θα δημιουργήσουμε πιο πολλέ ευκαιρίε για αυτέ τι μακροπρόθεσμε επενδύσει, τι οποίε ανυπομονείτε και εσεί να δείτε. Συμφωνώ μαζί σα απόλυτα ότι το σχεδίο Juncker των 315 εκατομμυρίων, είναι ε, μία αρχή μόνο, ένα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο μέτρο. Η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών από τη φύση της είναι μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος στον Επιτροπό Χίλ. Δυστυχώς, από ό,τι μου λένε, θα πρέπει να κλείσουμε εδώ την ε, συνεδρίασή μας, γιατί πρέπει να φύγει, να πάει σε αεροδρόμιο, έχει πτήσει προς τη ΣΥΠΑ. Ο Επίτροπος ζητώ συγγνώμη, προ προς συναδέλφου που έπρεπε να έχουν πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερω Επιτροπέ Χίλ για την παρουσίασή σας εδώ σήμερα, για την πολύ καρποφόρα αυτή συζήτηση. Θα συνεχίσουμε ασφαλώ την συνεργασία μαζί σας για το φάκελο αυτό των, της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Παρακαλώ οι δημοσιογράφοι να φύγουν. Πρέπει να ξεκινήσουμε την ε, συνάντησή μας.

I welcome... Καλωσορίζω τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Γερούν Ντάισελμπλουμ, για τον ε, οικονομικό μας διάλογο. Όπως θα γνωρίζετε, ο οικονομικός μας διάλογος με το Eurogroup είναι ένα καθοριστικό εργαλείο για να για το διάλογο με το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι βασικό στοιχείο του ρόλου του Eurogroup στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. Και είναι και ένα στοιχείο του συνόλου της δημοκρατικής λογοδοσίας μας. Όπως ξέρετε, το Eurogroup είναι ένας πρωτότυπος ε, θεσμός που έχει ιδιαίτερο ρόλο στη συνθήκη. Δεν είναι νομοθετικού χαρακτήρα, αλλά είναι ζωτική σημασία του για την ε, διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Έχει πολύ σημαντικές αρμοδιότητες και βεβαίως μετά την ε, δημιουργία του πλαισίου των μηχανισμών σταθερότητας που είναι βασικό εργαλείο της διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ακόμα και αν μερικοί από αυτού του μηχανισμού έχουν χαρακτήρα διακυβερνητικό και πάλι το Eurogroup γίνεται ακόμη πιο σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει και μια παρακολούθηση, ένα δημοκρατικό έλεγχο, να υπάρχει ένα υπόλογο προ του πολίτε. Γι' αυτό λοιπόν στην Επιτροπή μα ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά και ευχαριστούμε τον πρόεδρο Ντάισελμπλουμ για την δέσμευσή του, ώστε να έχουμε συστηματικό διάλογο μαζί του στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπως θα ξέρετε, στις προτεραιότητές μας για τον οικονομικό διάλογο. Έχουμε τη γενική επισκόπηση του τι γίνεται στην Ευρωζώνη, ποια είναι η οικονομική της κατάσταση. Βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή για τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ούτως ή άλλως και βεβαίως είμαστε και στην καρδιά μια συζήτηση στρατηγικής σημασίας για να δούμε τι θα γίνει με το πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας. Είμαστε λοιπόν εδώ για να ακούσουμε τον πρόεδρο Μπλουμ για την όλη κατάσταση για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα, τι θα γίνει με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έβαλαν χθε οι ελληνικές αρχές και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και σας δίνω αυτή αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι στην ΕΚΟΝ. Πριν έρθω στην Ελλάδα. Θα ήθελα όμως ε, να αναφέρω κάποια ευρύτερα ζητήματα, αν μου επιτρέπετε, γιατί ε, δεν υπάρχει μόνη κατάσταση στην Ελλάδα. Έχουμε και άλλα στην Ισια Διάταξη. 1η Ιανουαρίου, όπω γνωρίζετε, η Λιθουανία έγινε το 19ο μέλο τη Ευρωζώνη. Η εισαγωγή του ευρώ είναι ένα επίτευγμα που το άξιζε η χώρα διότι ακολουθεί μια εντυπωσιακή ε, διαδικασία σύγκλησης με εντυπωσιακά αποτελέσματα οικονομικής προσαρμογής ε, με την έξοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης. Ε, έγινε πολύ ομαλά η μετάβαση στο ευρώ και υπάρχει και μεγάλη υποστήριξη για τον νεονόμισμα από την κοινή γνώμη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προβλέψεις. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντηση του Eurogroup συζητήσαμε τις προβλέψεις για την Ευρωζώνη. Υπάρχουν λόγοι για συγκρατημένη αισιοδοξία. Η Επιτροπή περιμένει η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη να φτάσει στο 1,3% το 2015 και να αυξηθεί σε 1,9% τουλάχιστον αυτές είναι εκτιμήσεις για το 2016 η εγχώρια ζήτηση έχει σημειώσει άνοδο. Η μείωση δε των τιμών της ενέργειας σε συνεργασία με την ε, ε, θετική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, επηρεάζει τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτά είναι οι καλές ειδήσει. Πρέπει να είμαστε όμως ρεαλιστές. Οι υποστηρικτικές νομισματικές πολιτικές δεν μπορούν μόνες τους να ε, εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αυτό δεν μπορεί να το καταπετύχει και μόνο η μείωση των τιμών του πετρελαίου. Θέλουμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, άρα πρέπει να επεξεργαστούμε τις δομικές μεταρρυθμίσεις για να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα, παραγωγικότητα. Θέλουμε παραγωγικές επενδύσεις για να είναι πιο ανταγωνιστικές οι οικονομίες και βέβαια πρέπει να διατηρήσουμε την φορολογική ε, συνετή, φορολογική πολιτική και εποπτεία για να έχουμε ανάπτυξη. Και γι' αυτό βέβαια ξέρουμε ότι το προαπαιτούμενο είναι η ασφάλεια. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πρόοδο στους τομείς αυτούς ως Eurogroup η δημιουργία των κατάλληλων δροτικών πολιτικών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, ιδίως ε, εάν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί παραγωγικά η ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέλουμε να είναι πιο αποτελεσματικές οι αγορές εργασίας, ώστε οι άνεργοι να μπορέσουν να βρουν ε, δουλειά. Θα πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση των αγορών υπηρεσιών ε, και προϊόντων για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις, για να αυξηθεί ο ανταγωνισμό και να πάψει η κατάσταση με τα κλειστά επαγγέλματα. Και βέβαια πρέπει να βελτιώσουμε και, την ε, περίπτωση, και την, το φορολογικό άχρος να το μετατοπίσουμε από την εργασία. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ε, και ήδη έχουν ε, ξεκινήσει σε όλη την Ευρώπη. Είχαμε τις συστάσεις της Ευρωζώνης του 2014, συμφωνήσαμε ως Eurogroup επικοινών αρχών για να μειωθεί το φορολογικό άχθρο στην εργασία. Θα στρέψουμε την προσοχή μας ε, σε ορισμένε από αυτέ τι συστάσει ε, του Eurogroup στη διάρκεια τη χρονιά, ε, συνεργαζόμενοι στενά για τι πολιτικέ μα και για να θεσπίσουμε όπου είναι δυνατόν κάποιε κοινέ κατευθύνσει. Έρχομαι στι επενδύσει, φυσικά στο ECOFIN συνεχίζεται η δουλειά για το πρόγραμμα επενδύσεων και τη χρηματοδότηση πρωτοβουλία για την ανάπτυξη. Είναι σημαντικά αυτά γίνονται και στο Κοινοβούλιο πάρα πολύ σημαντικέ εργασίε προ αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να έχουμε βιώσιμα επενδυτικά προγράμματα και δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση που μπορεί να δώσει άμεσα αποτελέσματα. Πρέπει να βελτιώσουμε το επενδυτικό κλίμα και γι' αυτό δεν χρειάζονται μόνο δημόσια μέσα. Θα πρέπει και η εσωτερική αγορά να ενισχυθεί και να ολοκληρωθεί. Θέλουμε να εργαστούμε προς μια ανασκέφαλη αγορών. Έχουμε δε και το ψηφιακό θεματολόγιο, τα ενεργειακά δίκτυα. Όλα αυτά θα παράσχουν νέες επενδυτικέ ευκαιρίες. Σε ό,τι αφορά την φορολογική πολιτική, πολύ πρόοδο έχει επιτελεστεί. Γνωρίζετε ότι μειώθηκαν στην Ευρωζώνη τα ελλείμματα στο 2,6% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο έπεσαν το 2014 και η μείωση συνεχίζεται και προβλέπεται να είναι της τάξης του 2,4% κατά μέσο όρο πάντα για φέτος. Πάλι είναι υψηλά βέβαια, από μια έννοια. Χρειάζονται λοιπόν ε, προσπάθειες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ίσως ε, ύφεση, αλλά η πρόοδος είναι σταθερή προς το παρόν. Για δεύτερη χρονιά είχαμε ένα ειδικό Eurogroup ε, που έγινε το Δεκέμβριο για να θεωρήσει όλα τα δημοσιονομικά σχέδια. Δεν θεωρήσαμε ότι υπάρχει κάποιο από αυτά που δεν ε, συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα και τις χρεώσεις στο πλαίσιο του σχεδίου σταθερότητας, του Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι πάντως ε, και εμείς θέλουμε να τις ε, αντιμετωπίσουμε. Έγινε μια άσκηση αξιολόγηση από ομοτήμους και το Μάρτιο θα γίνει τελική, θα, τελική αξιολόγηση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά αυτές τις αναλύσεις. Να έρθω τώρα στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής ή επιτήρηση μετά την ολοκλήρωση προγράμματος. Ξεκινώ με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Είχαμε κάποιες αποστολές επιτήρησης που ολοκληρώθηκαν και στις δύο χώρες στα τέλη του 2014. Η Ιρλανδία συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο σε όλα τα μέτωπα, πολύ θετικέ εξελίξεις. 4,8% ανάπτυξη ήταν ε, τα ποσά της Ιρλανδίας το 2014 και η πρόληψη για το 2015 είναι 3,5%. Η ανάπτυξη ε, ε, μάλλον η απασχόληση σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο πέρυσι και αναμένεται η αύξηση να ε, διατηρηθεί και φέτος. Ε, στην Πορτογαλία το αίσθημα γενικά για την οικονομία, οικονομικές χρηματοπιστωτικές συνθήκες βελτιώνονται, έχουμε συνετές φορολογικές πολιτικές, διατηρίζεται οι μεταρρυθμίση, η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε, αυξάνεται η εξωτερική ζήτηση και η Κομισιόν προβλέπει ότι σταδιακά ε, η οικονομία και τα δημόσια οικονομικά της Πορτογαλίας ανακάμπτουν και σταδιακά μειώνεται και η ανεργία για την Κύπρο. Και αυτή έχει σημειώσει σταθερή πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματο. Είχαμε πρόοδο στο φορολογικό, στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και αναμένεται η κυπριακή οικονομία να επανέλθει στην ανάπτυξη το 2015. Όμως ε, η αναστολή ε, της ψήφης νομοθεσίας, ε, της νομοθεσίας για, τους, για τις αποκαλύψεις ε, τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, το λεγόμενο foreclosure, είναι κάτι αρνητικό γιατί είναι απαραίτητο ο νόμο αυτός στο πλαίσιο του προγράμματος και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έρχομαι στην Ελλάδα. Την προηγούμενη Πέμπτη, οι ελληνικέ αρχέ επισήμω ζήτησαν παράταση του προγράμματο που γνωστό είναι ως κύρια σύμβαση χρηματοδοτική διευκόλυνση, MFAFA, εμείς μπορούμε να το ονομάζουμε αυτό σύμβαση ή πρόγραμμα ε, ως πιο απλό και ζητήθηκε επίσης ε, και η περίοδος διαθεσιμότητας ε, των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χωματοψηφίας Σταθερότητας να παραμείνει στο μαξιλαράκι, αν θέλετε, του Ελληνικού Ταμείου Χωματοψηφίας σταθερότητα Για την πορεία μας από εδώ και πέρα συμφωνήσαμε την Παρασκευή. Θα σας αναφέρω τα βασικά στατικά. Θέλουμε ε, η Ελλάδα να έχει χρόνο παραπάνω για να μπορέσει να υλοποιήσει τους υφιστάμενους στόχους ε, της σύμβασης. Επίσης, ε, ζητώντας την παράταση, έκαναν ελληνικές αρχές και κάποιες, ανέλαβα κάποιες δεσμεύσεις μεταξύ αυτών. Να μην καταργήσουν μέτρα τα οποία ήδη έχουν ληφθεί και να απόσχουν από μονομερει ενέργειες που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους φορολογικούς, δημοσιονομικούς στόχου, την οικονομική ανάκαμψη και την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεσμεύτηκαν επίσης να τιμήσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις ε, προς όλους τους πιστωτές ε, και επίσης δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα για να έχουμε βιωσιμότητα του χρέου. σύμφωνα με τη δήλωση του Γιώργου το Νοέμβριο του 2012. Συμφωνούμε ε, ότι θα πρέπει να συνεργαστούν οι ελληνικέ αρχέ με το Eurogroup, με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το Θέσιο Νομισματικό Ταμείο για να γίνει καλύτερη χρήση τη ευελιξία. Και ε, αν είναι δυνατόν τα συμφωνημένα μέτρα να αντικαθισταθούν από άλλα που εκπληρώνουν του ίδιου στόχου, αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο τη ευελιξία αυτή. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει την ισχυρή της δέσμευση για ευρείες βαθιές διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, για βελτίωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της σταθερότητας, ανθεκτικότητας του σηματοπιστωτικού τομέα. Χθε παρουσίασε μια πρώτη λίστα μέτρων η Ελλάδα. Κάποιες εφημερίδες πάνω ότι δεν έγινε αυτό. Έγινε όμως, το επιβεβαιώνουμε και σήμερα θα γίνει αξιολόγηση από την Κομισιόν, την ΕΚΤ και το νιτάφ και ήδη θα ξέρουμε σήμερα, θα έχουμε μια πρώτη άποψη για το κατά πόσον είναι επαρκώς περιεκτικά αυτά τα μέτρα για να αποτελέσουν μια κανοποιητική αφετηρία. Με βάση τη Συμφωνία τη Παρασκευή, ε, τα κράτη-μέλη του Eurogroup ε, θα ξεκινήσουν τι απαραίτητε εθνικέ διαδικασίε για την τετράμινη παράταση τη σύμβαση και για τη διατήρηση αυτών των ομολόγων στο Ελληνικό Ταμείο. Οι ελληνικέ αρχέ στη συνέχεια θα ε, δώσουν περισσότερες πληροφορίες ε, σε σχέση με τα μέτρα τα οποία παρουσίασαν χθε και ελπίζουμε η συμφωνία με τα θεσμικά όργανα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου το αργότερο μόνο η έγκριση της ε, ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας ανθρώσης θα ε, επιτρέψει την εκταμείευση της τελικής ε, δόσης στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του Ταμείου Χροντοψικής Σταθερότητας και, των κερδών, και τη μεταφορά των κερδών στο πλαίσιο του προγράμματος των αγορών αξιογράφων. Τα, ταμεία, τα ομόλογα θα παραμείνουν στο ελληνικό ταμείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και κόστος ε, εξυγίανσης και θα απελευθερώνται, θα αποδεσμεύονται αυτά τα ομόλογα μόνο αν το ζητήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο νέος φορτικός μηχανισμός. Θέλουμε ουσιαστικά αυτό το πρώτο βήμα να ε, αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των πλευρών θέλουμε να μπει ξανά σε τροχιά η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, η ανάκαμψη. Και με την παράταση αυτή έχουμε χρόνο πλέον για να επεξεργαστούμε τη μελλοντική μας συνεργασία με την Ελλάδα και να ε, βρούμε αυτή την ε, περίοδο γέφυρα που χρειάζεται. Ε, αυτά τα κατάφεραν συμφωνήσεις Παρασκευής. Εδώ ολοκληρώνω και είμαι διαθέσιμος για Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Eurogroup και τώρα ξεκινάμε με τον γύρο ερωταπαντήσεων. Πρώτο ομιλητής είναι ο συντονιστή του ETP. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ντέσσελμπλουμ. σας καλωσορίζω και σας ε, ευχαριστώ για την ε, πολύ διαφανή άσκηση των καθηκόντων σε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα που είπατε ότι η ελληνική κυβέρνηση χωρίς καθυστέρηση παρουσίασε την λίστα, τον κατάλογο αυτό και με μεγάλη προσοχή χτες ε, διάβασα μια συνέντευξη του κ. Βαρουφάκη, του Υπουργού Βαρουφάκη στο CNN, ο οποίος είπε ότι δεν ήμασταν υπεύθυνοι εμείς για την καθυστέρηση. Το Eurogroup ζήτησε να τα καταθέσουμε αυτά την τρίτη το πρωί. Τι είναι λοιπόν, ποια είναι η άλλη αλήθεια. Θα ήθελα μια ανοιχτή απάντηση από πλευρά σας. Γιατί είπατε επίσης ότι ε, θα πρέπει να, υπάρξει εκ νέου εμπιστοσύνη. Η δική μου εντύπωση είναι ότι ιδιαίτερα στις τελευταίες εβδομάδες από την αρχή των καθηκόντων της θητείας της νέας, ευρωπαϊκής, της ελληνικής κυβέρνησης έχει χαθεί πολύ η εμπιστοσύνη. Πιστεύετε λοιπόν, ρωτώ, ότι είναι δυνατόν γρήγορα να αναξηθεί μια νέα εμπιστοσύνη, το οποίο θα ήταν απαραίτητα ασφαλώς. Και φυσικά μετά υπάρχει το ερώτημα του πώς σοβαρή είναι η ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα θέματα μεταρρυθμίσεων. Επί σειρά ετών το διαπιστώσαμε και είσαστε και πρόεδρος του Eurogroup, το ζήσατε λοιπόν στο πετσί σας. Ακούσαμε πολλές υποσχέσεις. Πόσο λοιπόν στα σοβαρά μπορούμε να πάρουμε τις εξαγγελίες για μεταρρυθμίσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, δεν υπήρξε καθυστέρηση. Δεν μπορώ λοιπόν να σας πω ποιος ευθύνεται για κάτι το οποίο δεν υπήρξε. Η ελληνική κυβέρνηση της είχε ζητηθεί. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν ε, έπρεπε να παρουσιάσει ένα κατάλογο προθέσεων ε, την ε, Δευτέρα και στις 11 και τα λοιπόν κατέφτασε στο δικό μου mailbox. Δεν υπήρξε καθυστέρηση. Έχει ζητηθεί πιο πολύ χρόνος. Είμαστε όμως στη σωστή τροχιά σε ό,τι αφορά τα θέματα χρονοδιαγράμματος. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Ρωτήσατε για θέματα εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να διευκρινίσουμε ότι τις πρώτες εβδομάδες μετά τις ελληνικές εκλογές υπήρξε διακύβευση πολλή εμπιστοσύνη μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά θεωρώ ότι αυτά που έγιναν την Παρασκευή ήταν ένα πρώτο βήμα προς την επαναφορά της εμπιστοσύνης αυτής. Η ερώτησή σα αφορά για το πόσο σοβαρή είναι η, Ευρωπαϊκή, η ελληνική κυβέρνηση για τι μεταρρυθμίσει. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρή. Αλλά είναι μια νέα ε, ελληνική κυβέρνηση με πολύ διαφορετικό όραμα. Θέλουν κάποιε αλλαγέ στις συμφωνίες λοιπόν. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα πετύχουν τους στόχους τους σε ό,τι αφορά την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την οικονομική ανάκαμψη, την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Αλλά η ευελιξία εντός του προγράμματος πάντα υπήρχε. Πάντα μιλούσαμε με τι κυβερνήσει, διαπραγματευόμασταν Ε, να αλλαγέ στο χρονοδιάγραμμα, αντικαθιστούσαμε μέτρα. Ακριβώ αυτό θέλει να κάνει η νέα ελληνική κυβέρνηση. Θα πρέπει να υπάρξει έντονη συνεργασία. Δεν μπορεί να υπάρξει μονομερή δήλωση ότι α, θα αλλάξουμε το μισό πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή συνεννόηση. Όσο τουλάχιστον θέλουν περαιτέρω χρηματοδότηση από την Ευρωζώνη. Αυτή είναι η προπόθεση. Είναι σοβαρή δεν πρόκειται να είναι απλό και εύκολο. Είναι ένα πρώτο βήμα αυτό μόνο. Αυτή η λίστα είναι ένα πρώτο βήμα, μια πρώτη ένδειξη για τις προ... μεταρρυθμίσεις που θέλουν να κάνουν, για τις αντικαταστάσεις που θέλουν να κάνουν, για αυτά που θέλουν να συνεχίσουν. Και ασφαλώς θα πάρει χρόνο το να υπησέλθουμε σε λεπτομέρειες, το να καταρτήσουμε μια νέα συμφωνία η οποία θα μας οδηγήσει πέρα από τους επόμενους τέσσερις μήνες. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος συντονιστή ε, ε, του Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ελίζα Ευχαριστούμε, για τα στοιχεία που μας δώσατε. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, οι απαντήσεις σας όταν η Επιτροπή ΕΚΟΝ σας προσκάλεσε να έρθετε και σας ρωτήσαμε πόσο είναι υπόλογη στον πρόεδρο του Eurogroup η Τρόικα. Και είπατε ότι ως πρόεδρος του Eurogroup δεν έχετε αρκετού συνεργάτε, προσωπικό ή ομάδε για να διαπραγματεύεστε εσεί απευθεία και να παρακολουθείτε τι λεπτομέρειε. Άρα ε, εμπιστεύεστε την αποτίμηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ε, περασμένη εβδομάδα στι συναντήσει του Eurogroup είδαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει υποβάλει μέσω του Επιτρόπου Μοσκοβισή προτάσει για το ελληνικό πρόγραμμα που ε, Έλλην Υπουργό Οικονομικών είπε ότι θα μπορούσε να προσυπογράψει. Όμω μετά αυτό ε, δεν έμεινε στο τραπέζι και έπεσε μια νέα πρόταση. Αυτό προκάλεσε εντάσει και υπήρχε κόστος στην εμπιστοσύνη και βεβαίω αυτό φάνηκε και στις χρηματοπιστωτικές αγορές με αυτή τη μεγάλη, τη μακρά καθυστέρηση. Τι έγινε, Ποιο ευθύνεται, ποιο χειρίζεται την ημερήσια διάταξη, τι έγινε με τη δική σα σχέση εμπιστοσύνη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη έχει να κάνει με την παρακολούθηση του θέματο. Έχετε ήδη σε εξέλιξη διαπραγματεύσει και πρέπει να σταθεροποιηθεί το κλίμα. Κατά πόσο συμμερίζεστε τι δηλώσεις, Ντράγκη, που λέει ότι θα διαφυλαχθεί η Ευρωζώνη ό,τι και αν χρειαστεί να γίνει και επίσης την εγγύηση του κυρίου Γιούνκερ ότι δεν θα υπάρξει έξοδος της Ελλάδας. Αυτό παραμένει μια σταθερά στις προτεραιότητές σας και ποιο είναι το πνεύμα των διαπραγματεύσεων που πρέπει να συνεχιστούν και με τη νέο κατάλογο διευθυντικών μεταρρυθμίσεων που προτάθηκαν. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον, και τα έχω ξαναπεί αυτά, ε, το έργο των ε, θεσμικών οργάνων είναι συμβουλευτικό ως προς το Eurogroup. Είναι όντως μικρή ομάδα συνεργατών μου και είναι αδύνατο να κάνουν τη δουλειά που και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορούν να κάνουν από κοινού για αυτά τα προγράμματα. Αλλά ε, είναι δική μας η απόφαση. Όταν λένε όλοι ότι φταίει η Τρόικα, εγώ λέω ότι κανονικά το Eurogroup θα πρέπει να κατηγορήσουν. Απλώς ε, έτσι, πηγαίνουν τα, ε, ε, έτσι καθορίζεται πώς θα πάει το χρήμα από τα ευρωπαϊκά ταμεία προς αυτούς που το χρειάζονται. Τώρα για τις προτάσεις του Επιτρόπου. Υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και των υπολείπων των μελών του Eurogroup σε μια-δυο συναντήσεις που ήταν ε, απαραίτητες για να καταλήξουμε σε μια λύση που θα μπορούσε να δεχτεί και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι υπόλοιποι 18 υπουργοί. Νομίζω λοιπόν ότι ο χρόνος χρειαζόταν. Αν δούμε τι έγινε το τελευταίο 15ήμερο, ήταν απαραίτητο αυτό για την ελληνική κυβέρνηση για να συνειδητοποιήσει ποια ήταν ακριβώς η κατάσταση της Ελλάδας και οικονομικός και δημοσιονομικός και πολιτικό. Και έπρεπε να συζητήσουμε στον κύριο Γκρουπ πώ θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ή να μην αλλάξουμε, ε, να τροποποιήσουμε τι υπάρχουσε συμφωνίε. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό. Δεν θέλω να επεκταθώ και να ε, επαστρέψω στο, στην πορεία αυτών των προτάσεων. Ήταν απαραίτητη διαδικασία και από πολιτική άποψη είδαμε και την ουσία των προγραμμάτων. Συμφωνώ κατά πολύ και με τον Μάριο Ντράγκη και με τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, το Brexit, η έξοδο τη Ελλάδα από την Ευρωζώνη, καν συζητιέται. Δεν έχουμε καν προετοιμάσει του εαυτού μα γι' αυτό, ούτε σκέψει. Η δική μου σταθερά είναι ότι θα πρέπει το Euro, η Ευρωζώνη να παραμείνει ενωμένη, ανθεκτική ε, και στα δύσκολα. Πολλέ φορέ υπάρχουν δυσκολίε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα, αλλά πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Αυτή είναι η δική μου θέση και η δική μου υπόσχεση. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, ο κύριος Στέρχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω και εγώ επί του ιδίου θέματος, κύριε Μετά τις ε, διάφορες ε, τοποθετήσεις σας τώρα υπήρξαν φήμες για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαν να το σκέφτηκε όπως και κάποια κράτη-μέλη που φαίνεται να έχουν προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Με τις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να μην υπάρχει τέτοια άμεση προοπτική. Όμως κάθε εβδομάδα έχουμε και καινούργια στοιχεία, νέες εξελίξεις. Δεν ξέρουμε πώς θα σταθερεί η νέα κυβέρνηση για παράδειγμα. Οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας. Υπάρχει η, δυνατό, η περίπτωση Brexit Γι' αυτό και νομική βεβαιότητα για το πώ θα φύγει ένα μέλος μέλο από την Ευρωζώνη χωρί να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν καλό αυτό να το γνωρίζουμε για τα ερχόμενα χρόνια κατά τη θητεία σα. Οπότε ε, η ερώτησή μου είναι εξή. Τι είδου πολιτικό, οικονομικό ή νομικό πλαίσιο μπορείτε να φανταστείτε να συζητιέτε στο Eurogroup ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αρνητικών πολλαπλών συνεπειών εφόσον μια χώρα βγει από την Ευρωζώνη. Γιατί κανονικά αυτή τη συζήτηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την παραγωνίσουμε σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Ξέρετε ότι η περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται από τις συνθήκες. Αλλά το λόγο έχει ο πρόεδρος του Eurogroup. Πολύ καλή απάντησή σας είπατε ότι πολλά κράτη-μέλη προετοιμάστηκαν. Εγώ άκουσα μία χώρα όπου οι διάφοροι υπουργοί συναντήθηκαν για να συζητήσουν μια πιθανότητα Brexit και ήταν ακριβώς η Βρετανική. Αυτό το άκουσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όπως θα ξέρετε η Βρετανία το ή ακόμα δεν είναι μέλη του Eurogroup δεν συζητήθηκε και αυτό αποδεικνύει την ε, σαφή πολιτική μας αφοσίωση και υπόσχεση να παραμείνει ε, άθικτη η Ευρωζώνη, σώα και ενωμένη και νομίζω ότι αν οι πολιτικοί θύνοντες δεν έχουν τέτοια αφοσίωση, αυτό θα έδινε πολύ περίεργα μηνύματα για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση που έχουμε οικοδομήσει. Τι εμπιστοσύνη θα υπήρχε. Εγώ Πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε. Υπάρχει έδαφο και κοινό έδαφο συνεννόηση. Αυτό κάνουμε εδώ και καιρό. Αυτό κάνουμε την τελευταία διετία. Συνεχίζουμε και ενισχύουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τι κοινέ μα δεσμεύσει. Αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι είναι σκόπιμο να επιστρέφουμε διαρκώ στην δυνατότητα, την πιθανότητα ε, τη εξόδου χωρών από την Ευρωζώνη. Έχουμε διοικητεύσει πάρα πολύ κεφάλαιο και κυρίω πολιτικό, πολλή δουλειά για να γίνει ε, ισχυρή αυτή η Ένωση. Και πρέπει να παραμείνουμε σε αυτήν την άγουσα. Πολλές χώρες είναι ακόμη ευάλωτες. Η απάντηση για τις χώρες αυτές δεν είναι να βγουν από την Ευρωζώνη, αλλά ε, ούτε απλώς να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε την Ευρωζώνη. Το θέμα είναι αν με την Ευρωζώνη και με τους Ευρωπαίους εταίρους τους μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες και τα ευάλωτα σημεία που υπάρχουν ε, στις οικονομίες τους, στις κυβερνήσεις, και την κυβερνητική του δομή και ούτω καθεξής. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τα φέρουμε εις πέρας. Ναι, για να αντιτυπώσω την ερώτησή μου. Ήμασταν πολύ κοντά σε μια κατάσταση όπου είχαμε μια κυβέρνηση πριν από τις εκλογές, είχε υποσχεθεί να αλλάξει την πολιτική και τώρα φαίνεται ότι παίρνουν πίσω τις υποσχέσεις που έκαναν στο λαό τους. Τι θα γίνει όμως αν η κυβέρνηση αυτή δεν πάρει πίσω τις υποσχέσεις της για τους ε, νέους κανόνες ή για την έξοδο. Τι θα κάνετε τότε, αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν ε, ξεκίνησα την πολιτική για να κάνω εικασίες ή για να προετοιμάζομαι για το χειρότερο. Μπήκα στην πολιτική για να προετοιμάζομαι για το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμώ, επιθυμούμε. Τι επιθυμούμε λοιπόν. το ίδιο που θέλει και η νέα ελληνική κυβέρνηση. Να έχει η Ελλάδα τη θέση της στην Ευρωζώνη υπάρχει ισχυρή υποστήριξη στο μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού, λαού για την Ευρωζώνη. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους, πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στον δημόσιο και ειδικό τομέα στην οικονομία της Ελλάδας. Αυτό θα είναι δύσκολο, θα πάρει χρόνο. Θα, ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει αποφασιστικότητα των πολιτικών και στην Ελλάδα κυρίως, αλλά και στο Eurogroup. Και γι' αυτό εργαζόμαστε. Thank you. Σας ευχαριστώ, Ρόγιο Πρόεδρος. Από πλευρά της Άλντες, η κόρα φανιουάζουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα μιλήσω στα Ολλανδικά. Και γιατί αυτό είναι δυνατόν με τον κύριο Ντέισελμπλουμ. Καλώ όρισε, Γερούν, και πάλι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε άλλο ένα έργο στο ελληνικό δράμα. Δεν θα είναι και το τελευταίο, δυστυχώ. Οι μεταρρυθμίσει δεν έχουν γίνει ακόμα οι μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα Θέλω να κάνω μια ερώτηση όμως για τις μεταρρυθμίσεις αυτές, γιατί ο Μάριο Ντράγκη με πολύ μεγάλη σαφήνεια είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποίησε το τελευταίο χαρτί διάσωσης ε, της οικονομικής πολιτικής και τώρα εξαρτάται και επαφίεται στα κρατή μέλη της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης να καταστεί ανταγωνιστική η Ευρώπη και να περάσουν οι μεταρρυθμίσεις. Εσείς ως επικεφαλής του Eurogroup πώς θα φροντίσετε οι χώρε πραγματικά να περάσουν τις μεταρρυθμίσει αυτέ. Γιατί κοιτώντα το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, έχουμε ανακαλύψει πιο πολύ σταθερότητα. Μπορώ λοιπόν να υποθέσω ότι όπως έχει διαμορφωθεί έχουμε εξαντλήσει τα όρια της σταθεροποίησης. Ξέρουμε λοιπόν που βρισκόμαστε, αυτό είναι το πακέτο, αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα πετύχουμε αυτά. Φαίνεται ότι η Γαλλία έδωσε στον εαυτό τη άλλη μια νέα παράταση. Πώ μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μεταρρυθμίσεων των διαρθρωτικών, Γιατί θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τη μοναδική σανίδα σωτηρίας για την αντικανοστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σα. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο και βάση για αισιοδοξία. Προσεκτικά βέβαια ο ΑΣΑ δημοσίευσε μία μελέτη πριν από κάποιους ε, μια μελέτη για την ε, πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Υπάρχει σαφής πρόοδος λοιπόν. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν ε, προχωρήσει στις χώρες προγραμμάτων, στα πλαίσια των προγραμμάτων, αλλά και στις βαλτικές χώρες για παράδειγμα. Και στη δική μου τη χώρα προωθούμε μια ισχυρή ατζέντα μεταρρυθμίσεων. Αυτό λοιπόν ε, εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη και αντιμετωπίζει κάποια από τα πιο κρίσιμα και βασικά θεμελιώδη προβλήματα που έχουμε. Και σε κάποιες περιπτώσεις το νομικό το σύστημα το ίδιο απειλεί τις επενδύσεις. Όλα τα ζητήματα λοιπόν αυτά αντιμετωπίζονται και στη Γαλλία όπως αναφέρεται Ο ΑΣΕ και στην Γαλλία κατέδειξε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αγορά εργασίας και σε άλλες μεταρρυθμίσεις. Και τις τελευταίες ημέρες γίνονται ακόμα πιο πολλές εξελίξεις και μεγαλύτερη πρόοδος στη Γαλλία. Πώς θα το πετύχουμε αυτό και πώς θα έχουμε πιο πολύ μόχλευση στην ίδια τη διαδικασία. Έχουμε πολύ μόχλευση στην παρούσα φάση, στην χρηματοπιστωτική πτυχή. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη μόχλευση και επιρροή σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Εργαζόμαστε για να υπάρξει πιο μεγάλο συντονισμό στο Eurogroup βάζοντα διαφόρων ειδών μεταρρυθμίσεις στην ατζέντα, κοιτώντα πώ γίνονται τα πράγματα στις διάφορες χώρες, συγκρίνοντας, αναπτύσσοντας βέλτιστες πρακτικές, αναπτύσσοντας πρότυπα για τις χώρες, φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερω. Επίσης υπήρξε ένα έγγραφο ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 1,5-2 χρόνια νομίζω ότι υπήρξε μία έκκληση να υπάρξει σύνδεση μεταξύ όσων γίνονται στις μεταρρυθμίσεις στο χρηματιστικό κλάδο, γιατί φυσικά υπάρχει και μακροπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος αντίκτυπος στην πλευρά του προϋπολογισμού. Γιατί, για παράδειγμα, το γεγονό ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα τη υγειονομική περίθαλψη έχει αντίκτυπο χρηματοπιστωτικό απαλύνει τι χρηματοπιστωτικές πιέσει. Στο προληπτικό λοιπόν σκέλο του συμφώνου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται, να επιτρέψουμε στι χώρε να πετύχουν του στόχου του αν πετύχουν και στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει λοιπόν στον κλάδο των μεταρρυθμίσεων να κοιτάξουμε να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τι χώρε να το πετύχουν. Αλλά συμφορώ απόλυτα μαζί σα, χρειάζονται διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. Είναι διαφορετικέ οι μεταρρυθμίσει οι διαφορετικέ που χρειάζονται σε κάθε χώρα. Θα πρέπει με ευφυή τρόπο να περνάνε. Με βαθμίο, σταδιακό τρόπο σε κάποιε περιπτώσει, για να απαλύνουν ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο. Είναι κρίσιμη σημασία να πετύχουμε ανταγωνιστικότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε υψηλό επίπεδο μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα από πλευρά τη ΓΚΟΕ ο κ. Παπαδημούλη. Κύριε Ντάισεμπλουμ, σα καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν λίγο διάβασα το πρώτο σχόλιο της Κομισιόν για τη λίστα μεταρρυθμίσεων που έγκαιρα κατατέθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Την χαρακτηρίζει επαρκώς περιεκτική και επίσης προσθέτει ότι η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυμένη από την ισχυρή δέσμευση της νέας ελληνικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Συμμερίζεστε αυτό το σχόλιο και εσείς προσωπικά που την έχετε δει. Θα ήθελα να καθησυχάσω τους δύο συναδέλφους των Γερμανών χριστιανοδημοκρατών και των Βρετανών συντηρητικών ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι και πολύ σοβαρή και πολύ σταθερή. Έχει την υποστήριξη του 80% των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, στις συζητήσεις που διεξάγονται και οι Έλληνες πολίτες υποστηρίζουν με ποσοστό 80% τη συμμετοχή στο ευρώ και δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνο Brexit. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα, κύριε Ντάισεμπλουμ. Το πρώτο, σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου του 2012, που και εσείς μνημονεύσατε, το Eurogroup δεσμεύεται από τη στιγμή που ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός σημειώσει πρωτογενή πλεονάσματα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα απομείωσης του ελληνικού χρέους χωρίς επιβάρηση φυσικά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Υπάρχουν προτάσεις από το Ινστιτούτο Μπρούγκελ σχετικές που έχουν κατατεθεί. Πότε σκοπεύει το Eurogroup να συζητήσει και να εφαρμόσει σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές τέτοια μέτρα. Και το δεύτερο, ξέρετε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα που τελειώνει προκάλεσε ύφεση 25% στην ελληνική οικονομία και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση πάνω από 25% ανεργία, 2,5 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από τα όρια της φτώχειας ζουν, 9 στους 10 Έλληνες ανέργους δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ επίδομα ανεργίας. Στην ανακοίνωση της Παρασκευής έχετε σημειώσει κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσματα. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θέλει πρωτογενή πλεονάσματα, θέλει νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, αλλά έχει ζητήσει μια αναπροσαρμογή ρεαλιστική προ τα κάτω των πρωτογενών πλεονασμάτων που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, που είναι 3 και 4,5% εξωπραγματικά. Πότε σκοπεύετε να κάνετε συγκεκριμένη τη λέξη appropriate, προκειμένου να ενισχυθεί μια δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Thank you very ε, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Κατά πρώτα να ρωτήσω αν συμβαίνει η αποτίμηση της Κομισιόν των πρώτων αυτών ελληνικών προτάσεων. Θα έλεγα ότι πρέπει τα τρία θεσμικά όργανα όταν να μας δώσουν κάποιες συμβουλές και αν είναι και τρεις θετικές, οι τρεις τοποθετήσεις θα έχουμε μια συνδεξιτή που για να ενημερωθούμε μεταξύ υπουργών θα λάβουμε γνώση και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Η διαδικασία τη βλέπω θετικά και πιστεύω ότι θα προχωρήσει. Πολλά όμω απομένουν να γίνουν από, από την πλήρη απάντηση. Μετά με ρωτήσατε τι θα κάνουμε με την λιωσιμότητα του χρέου. Και μιλήσατε για τι 12 Νοεμβρίου και τη σχετική συμφωνία στο Eurogroup και τι δηλώσει του για το 2012. Ε, εδώ, όταν αναφέρονται όλοι σε αυτό, μιλούν για ένα μόνο από τα κριτήρια. Όμως, τα κριτήρια ήταν πολλά. Το Eurogroup μπορούσε να σκεφτεί αν χρειαζόταν το τι θα γίνει με την δεσμότητα του χρέους το 2022 και αν τότε θα ε, πρέπει να αναλυθούν τα μέτρα για τη βιωσιμότητα του χρέου. Και βλέποντα αν έχει πρωτογενέ πλέον η Ελλάδα. Εάν έχει ε, καλύψει όλε τι δημιουργίε του προγράμματο, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Και νομίζω αυτά ήταν τα λόγια που υπόθηκαν. Το Eurogroup θα λάβει υπόψη και θα σκεφτεί έχουν δηλαδή υπάρξει θέμα βιωσιμότητα. Και ε, με την προπόθεση ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει όλε τι υποχρεώσει και όλε οι ε, υποσχέσει τη έχουν έρθει ει πέρα ε, επιτυχώ με μια πέμπτη αποτίμηση. Και μετά θα βλέπαμε τι είδου μέτρα πρέπει να αναλυθούν. Εάν λοιπόν αναφέρεστε σε αυτή τη δήλωση, μην ξεχνάτε τα υπόλοιπα τμήματά τη και απομονώνετε ένα από τα κριτήρια. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε βάσει τη παράταση του τετραμήνου εφόσον κάτι που θα επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να εκπληρώσει τι υποχρεώσει. τη. Εφόσον αυτό γίνει, τότε θα ολοκληρωθεί η περίοδο του προγράμματο. θα γίνει μια νέα ανάλυση και εξέταση τη βιωσιμότητας του χρέου και τότε θα δούμε τι επιπλέον, τι πρόσθετα μέτρα, εφόσον χρειάζεται, μπορούμε να αναλάβουμε ή να Νομίζω αυτέ ήταν οι ερωτήσεις Ναι, και εδώ καλό θα ήταν να διαβάσετε και την υπόλοιπη δήλωση. Λέει το δέον πρωτογενές έλλειμμα. Ε, πλέον, συγγνώμη. Και αναφέρεστε και πάλι στι δηλώσει του Νοεμβρίου 2012. Εκεί είχαμε καταλήξει σε μια συμφωνία για προσαρμογή του δεύτερου προγράμματος επειδή είχαμε καλύτερους αριθμούς για το πρωτογενές ε, ε, έλλειμμα ήδη τρία φέτο και 4,5 λέγαμε για το χρόνο. Τώρα αυτό είναι δέον και σκόπιμο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ε, στα τέλη τη περασμένη χρονιά η ελληνική οικονομία ε, βρέθηκε σε μια στάση. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει φέτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πρώτον θα αποτιμήσει αν οι δημοσιονομικοί στόχοι και οι προθεσμίε στηρίχθηκαν. Εάν δηλαδή η αύξηση του πρωτογενού πλεονάσματο είναι ακόμη εφικτά ε, λόγω των οικονομικών συνθήκων. Αυτό διαφέρει από να λέει μια κυβέρνηση ότι τώρα δεν θα σεβαστούμε πλέον καν αυτού του στόχου. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται μόνο με Με άλλα λόγια, εάν οι οικονομικέ προποθέσει μα δείξουν ότι υπάρχει περιθώριο, οι δημοσιονομικοί στόχοι μπορεί να προσαρμοστούν εντό των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Κάτι που ήδη έχει γίνει στο παρελθόν. Αλλά δεν μπορεί να είναι μια μονομερή απόφαση τη ε, ενδιαφερόμενη κυβέρνηση που να λέει πλέον δεν έχουμε δεσμεύσει, δεν έχουμε στόχου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.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 λέτε ότι επιβάλαμε συμφωνία στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση δεν το κάναμε αυτό. Αν η ελληνική κυβέρνηση είχε πει δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα πια, δεν θέλουμε αυτού του είδου τη συνεργασία πια, θα ήταν μια επιλογή κι αυτή. Αυτό το οποίο έγινε τώρα ήταν το εξή. Είπαμε, ακούστε, υπάρχει ένα πρόγραμμα ακόμη, α προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε, θα επιτρέψουμε όμω ευελιξία ε, πλέον στο πρόγραμμα και μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να την χρησιμοποιήσει αυτή την ευελιξία και να βάλει τη δική τη πολιτική φραγίδα στο πρόγραμμα. Και αν σεβαστεί η ελληνική κυβέρνηση, που είναι και προ το κοινό ε, συμφέρον το επαναλαμβάνω, του βασικού στόχου, δηλαδή βιωσιμότητα δημοσίων οικονομικών, οικονομική ανάκαμψη, σταθερότητα χρηματοπιστωτικού τομέα, αν δεχθούν και ε, σεβαστούν αυτού του βασικού στόχου, μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματο πολλέ αλλαγέ. Πολλή δουλειά έχουμε μπροστά μα. Θα πρέπει να δούμε τα συγκεκριμένα προγράμματα βέβαια και μέτρα και να τα μελετήσουμε. Έχουμε λοιπόν ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα. Ελπίζουμε να είναι πριν τα τέλη Απριλίου. Και σε από το δεύτερο ερώτημά σα που ουσιαστικά με ρωτάτε αν έχουμε αρκετό χρόνο δεδομένη τη χρηματοπιστωτική και χρηματοοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, θα σα απαντήσω ότι όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν πρέπει να χαθεί ε, χρόνο και πρέπει να περάσουμε στι απαιτούμενε προσαρμογέ, οποίε ε, ζητά η ελληνική κυβέρνηση, τι θέλει, αλλά μέσα στο εξάμενο πρόγραμμα. Θέλουμε να υπάρξει συμφωνία για να παραμείνει αυτό το πακέτο, να έχουμε ένα ισχυρό καλό πρόγραμμα και να ε, περάσουμε στην πράξη. Και με τα βήματα που θα γίνονται σιγά μπορούμε να παρέχουμε και χρηματοδότηση στην ελληνική κυβέρνηση. Πάντοτε έτσι εργαστήκαμε και καλά ε, λειτουργήσε αυτό το σύστημα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να μην χάνουμε χρόνο. Ας περάσουμε στις πράξεις. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα από πλευρά του Διευθυντή, ο Μάρκο Βάλλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα Ευχαριστώ, να

Ε, τελικά βρεθήκαμε με αυτό το αποτέλεσμα. Ε, ήθελα λοιπόν να σας ήθελα που αποδείξατε ότι υπάρχει μια τεχνοκρατική δικτατορία εδώ. Ε, αυτό επίση θα ενισχύσει και τον ευρωσκεπτικισμό και όσου δεν πιστεύουν σε αυτή την πραγματικότητα για τους πρόοδου τη στιγμή που το μόνο που έχετε είναι αριθμητικά στοιχεία και παραμέτρους. Ενώ δείχνουν τα στοιχεία Λουξεμβούργου ότι έχουμε απόλυτη δημοσιονομική ανομοιογένεια, ότι τα τελευταία αυτά χρόνια δεν έχουν προσφέρει τίποτε από άποψη πολιτικών στο Συμβούλιο. Υπάρχει κλίμα. Δεν προχωράει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πραγματικά είμαστε τελείω ετερογενεί. Και υπάρχουν μιλούσα για ρήξη την Ευρωπαϊκή ε, στην Ευρωζώνη ε, τα αποτελέσματα από τις ε, εκλογές. Ο Ντράγκη έχει πάρει κάποια μέτρα προετοιμαζόμαστε για Brexit, σε καμία περίπτωση, αλλά για την οικονομική ανάκαμψη, την περαιτέρω οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης, ε, που θα περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Θα ήθελα να πω, και θα είμαι πολύ σύντομος, κάποια πράγματα για το ενδεχόμενο επιστροφής μιας χώρας στο παλιό της νόμισμα, ότι αυτό θα ήταν ε, θετικά, θετικό από οικονομική Πρέπει να συνειδητοποιήσετε τι θα συνέβαινε αν μια χώρα γύριζε σε ένα πολύ πιο αδύναμο νόμισμα, αυτομάτως πολύ πιο αδύναμο από το ευρώ. Τι θα συνέβαινε αυτό και σε ό,τι αφορά την αξία ε, του χρέους που θα ήταν εντελώς πλέον ε, ε, μη βιώσιμο. Τι θα γινόταν και με τις αποταμιεύσεις των απλών ανθρώπων σε αυτή τη χώρα Ένας Ολλανδός οικονομολόγος είχε πει κάποια φορά ότι αν η υποτίμηση του νομίσματος είναι μια υγιής οικονομική ή νομισματική πολιτική, η Ζιμπάμπουε σήμερα θα έπρεπε να είναι πάμπλουτη ως χώρα. Άρα μακροπρόθεσμα είναι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας πολιτικής, αλλά μακροπρόθεσμες συνέπειες είναι πάρα πολύ αρνητικές. Κύριε Σαμονό, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε θεωρείται ότι η υποτίμηση του νομίσματος θα ήταν κάτι κακό. Πρέπει όμως να δούμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Αν τη στιγμή δηλαδή που αποκτήσει εκ νέου νομισματική ελευθερία η Ελλάδα με την Ελλάδα θα μπορούσε με την νομισματική της πολιτική ε, να καταφέρει να αποπληρώσει χωρίς κούρεμα το χρέος της, ε, υιοθετώντα κάποιες ε, νομισματικές ρυθμίσεις. Θα ήταν καλύτερο από το να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Ε, Όχι, δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι αυτό που θα βοηθούσε πραγματικά ε, την Ελλάδα είναι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Αυτό που γίνεται τώρα, αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε τώρα. Δηλαδή θέλουμε να βοηθήσουμε να γίνει πιο ισχυρά οικονομική Ελλάδα. Οι κρατικές υπηρεσίες ε, να είναι καλύτερες, η φορολογία να είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο και να είναι πολύ πιο δίκαιη η φορολόγηση, πιο αποτελεσματική ε, η φορολογία. Αυτά θα είναι τα κρίσιμα κατά με για την ανάκαμψη της Ελλάδας. Οι προτάσεις σας δυστυχώς φοβούμαι ότι μόνο θα αποσταθεροποιούσαν την κατάσταση. Πρόεδρος, ο κύριος, ε, ή μάλλον η Έστερ Ντελάνγκ από ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να, θα μιλήσω και εγώ στα Ολλανδικά, αν και φαντάζομαι δυστυχώς ε, το... η απάντηση θα είναι στα Αγγλικά. Σας ε, συγχωρώ, επίσης, είστε Πρόεδρος του Eurogroup. Δύο παρατηρήσεις έγιναν πολλέ παρατηρήσεις για την προηγούμενη εβδομάδα και για την επόμενη ε, περίοδο των τεσσάρων μηνών. Θα ήθελα να δω τι θα γίνει μετά τους τέσσερις μήνες. Έχουμε αγοράσει χρόνο, έχουμε εξαγοράσει χρόνο, Όντω, Μετά από τέσσερις μήνες όμως θα έχουμε και πάλι την ίδια συζήτηση. Εξίσου στεναρή. Ο πρόεδρο του Eurogroup τι ρόλο προβλέπει για τους θεσμικούς ε, φορείς που έχουν κάνει τόσα δάνεια προς την, προς την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το καθεξής. Όσο οι χώρες έχουν χρέη, θα πρέπει να εμπλέκονται οι θεσμοί αυτοί. Πώς μπορούμε λοιπόν να δώσουμε μορφή σε αυτή τη συμμετοχή. Δεύτερη ερώτηση. Μιλάμε πάρα πολύ για την Ελλάδα και δικαίω, γιατί έχουν συμβεί πολλά. Αλλά μήπως αυτό μας αποσπά την προσοχή από αυτά που συμβαίνουν στις άλλες χώρες. Πολύ θετική η αξιολόγηση των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων είσαστε για τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν συμφωνώ απαραίτητα, αλλά τουλάχιστον πρόκειται για ευθαπτικές μεταρρυθμίσεις, κοιτώντα τις ελλείψεις, τα ελλείμματα προϋπολογισμού, κοιτώντα τις πρωτοβουλίες και τις φιλοδοξίες του 2012 και το τι ακούμε τώρα από τη Γαλλία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να δείσουμε και άλλη παράταση για να φτάσουμε τον στόχο του 3% το 2018. Αυτές είναι οι φήμες που ακούγονται. Για πείτε μας λοιπόν πόσο ευκταίο θεωρείτε ότι είναι εκ νέου μια μεγάλη χώρα να την δώσουμε ίσως και υπερβολική ευελιξία. Μήπως είναι επικίνδυνο το προηγούμενο αυτό. Και μια Ολλανδική απορία, με παροιμία που άκουσα στο ραδιόφωνο. Ε, ίδια μέτρα και ίσα σταθμά ουσιαστικά. Αυτό θα έπρεπε να ισχύει και για τη Γαλλία. Ευχαριστώ κύριε Ντελάγκα και θα απαντήσω στα αγγλικά όντω. Καταρχάς, η περίοδος μετά τους τέσσερις μήνες. Οι τέσσερις μήνες θα μας επιτρέψουν δύο πράγματα. Να ολοκληρώσουμε το τρέχον πρόγραμμα, να κάνουμε μια ανάλυση λεπτομερή και να δούμε ποιες προκλήσεις παραμένουν στην Ελλάδα. Και βάσει της ανάλυσης αυτής θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε για περαιτέρω συνεργασία και υποστήριξη για την ελληνική κυβέρνηση. Πάντα λέγαμε στο Eurogroup ότι αν η Ελλάδα δεσμευτεί προς το πρόγραμμα και κάνει ό,τι πρέπει για να πετύχει τους στόχους, εμείς από πλευράς της Eurogroup του Eurogroup είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την περίοδο των τεσσάρων μηνών. Μετά τον Ιούνιο θα δούμε τι θα γίνει. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Τα θεσμικά όργανα θα συνεχίσουν να εμπλέκονται και να συμμετέχουν πολύ απλά γιατί έχουν ε, έντονα συμφέροντα. Το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα του 2016. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Ούτε σε τέσσερις μήνες θα έχει ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσει αν η Ελλάδα δεσμευτεί προς το πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα θεσμικά όργανα, ακόμα και αν δεν υπάρξει πρόγραμμα μετέπειτα ή συμφωνία μετέπειτα, follow-up. Και πάλι θα υπάρξει εποπτεία μετά τη λήξη του προγράμματος λόγω των μεγάλων συμφερόντων που σημαίνουν τα ε, δάνεια προς την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες χώρες που έχουν ολοκληρώσει προγράμματα, το ίδιο θα συμβεί και στην Ελλάδα αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε επιπλέον υποστήριξη για την περίοδο μετά το καλοκαίρι. Για τη Γαλλία τώρα. Ξέρετε ποια είναι η θέση μου. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με το μέγεθο τη χώρα η αντιμετώπιση τη κάθε χώρα. Δεν έχει σχέση αν είναι μικρή ή μεγάλη. Η Κομισιόν έχει δώσει και στον εαυτό τη και στην Γαλλία πιο πολύ χρόνο για να εξετάσει τα αριθμητικά στοιχεία, για να λάβει πιο πολλά μέτρα, για να προετοιμάσει πιο πολλέ προτάσει. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον όλες οι προτάσεις έχουν κατατεθεί ήδη. Θα τις αξιολογήσει στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας κάνει την σχετική έκθεση αρχές Μαρτίου. Ασφαλώς και είναι κρίσιμη σημασία για την αξιοπιστία όλου του χρηματοπιστικού συμφώνου να δεσμευτεί η Γαλλία για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Είπατε ότι ήμουν πάρα πολύ θετικό και αισιόδοξο. Εγώ απλά ανάφερα είπε η μελέτη του ΑΣΕ. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό μια μεγάλη οικονομία στην καρδιά της Ευρώπης να ανακάμψει. Και θεωρώ ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, η Εύα εφόσον η Ευρώπη και η Ελλάδα βρισκόνται στο επίκεντρο της προσοχής και το Eurogroup δυστυχώς επιμένει στη λιτότητα και αυτό μας είναι γνωστό. Κάποιοι θεωρούν ότι 30% ανεργία σημαίνει επιτυχημένα αποτελέσματα. Όμως η λιτότητα και πάλι αφισβητείται και μάλιστα ηχηρά. Τη στιγμή λοιπόν που οι διαδοτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα με τους μακροπρόθεσμου προσανατολισμούς και την φερεγγιότητα της χώρας, αυτά κάνουν τη ρευστότητα κάτι που μπορεί να γίνει πραγματικότητα και αυτό θα σκότωνε αμέσω την οικονομία. Ε, η ερώτησή μου λοιπόν έχει να κάνει με αυτό το σημείο. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προγραμματίσει μετά την δίμηνη τεχνική παράταση του προγράμματος τη μετάβαση σε μια ε, ε, δημοσιονομική γραμμή πρόληψης, η CCL. Τώρα με την νέα κυβέρνηση και την απόφαση να παραταθεί το πρόγραμμα από το Eurogroup. Υπάρχει τον Ιούλιο αυτή η πρόβλεψη για μια νέα γραμμή προφύλαξης ε, ή τέλο πάντων για ένα άλλο πρόγραμμα που ίσω θα περιλαμβάνει κάποιο νέο δάνειο. Πότε πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα πάρει τι επόμενε δόσει για το 2014. Διότι μέχρι τότε δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, ιδέες για το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες του Μαρτίου, λόγου χάρη. Η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε να καλυφθούν από το ELA, από τα ομόλογα της ελληνικής κυβέρνησης που θα αγόραζαν οι ελληνικές, τράπεζε. Τι πιστεύετε για αυτή την πρόταση, είναι αποδεκτή. Και τρίτη ερώτηση. Η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε, εξ όσων γνωρίζω, δύο νομοθετικές προτάσεις. Μία για 100 για ένα πρόγραμμα με 100 δόσεις για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στην αποπλήρωση αποπληρωμή των φόρων τους και μία για την διεύρυνση της προστασίας εξυπηρέτησης, κάλυψης μάλλον των ε, ε, χρεωμένων οικοκυριών από τις ε, από τους πληστηριασμούς της Πιστεύω ότι τα δύο αυτά προγράμματα μπορεί να διατηρηθούν, να σταθούν ή θα τα κρίνει η Τρόικα μετά τον Απρίλιο. Ευχαριστώ στι συνομιλίε μα με την προηγούμενη κυβέρνηση βλέπαμε το μέλλον και συζητούσαμε την δυνατότητα να υπάρξει υποπροποθέσει ενισχυμένη δημοσιονομική γραμμή προφύλαξη. Αλλά με ε, κάποιες ε, εξ προϋποθέσεις. Τώρα αυτό εφικτό είναι πολύ νωρί για να το πούμε. Πρέπει όμω να καταλάβετε ότι για να μπορέσει να είναι επαρκή αυτή η δημοσιονομική γραμμή, μια χώρα πρέπει να έχει πρόσβαση στι αγορέ και να μπορεί καταρχήν να αυτοχρηματοδοτείται. Μόνον εάν αυτό ισχύει ή οι αγορές λόγω δικών τους τρευλώσεων δεν είναι προσβάσιμες, τότε υπάρχει αυτή η δημοσιονομική δικων του τρευλωσεων Είναι ένα εργαλείο προληπτικό βέβαια. Για την ερώτηση αν η Ελλάδα θα επιστρέψει στις αγορές σε τέσσερις μήνες, θα σας τα αφήσω να τα απαντήσετε μόνοι σας. Ρωτήσατε τι θα γίνει με τι υπόλοιπε δόσει του 2014. Οι πληρωμέ από το πρόγραμμα πάντοτε εξαρτώνται από την επιτέλεση προόδου στα πλαίσια του προγραμματο και επιτυχημενε αναθεωρήσεις και αποτιμησει Νομίζω η τελευταία αποτίμηση ήταν πριν πολύ καιρό. Εδώ και κάποιο καιρό λοιπόν δεν προβλέπονται πληρωμέ από το πρόγραμμα προ την Ελλάδα. Μόλις αρχίσει το πρόγραμμα και η νέα κυβέρνηση ε, αρχίσει να προωθεί μέτρα εντός του προγράμματος και εντός της συμφωνίας, τότε μπορούμε να ξαναδούμε τις αποτιμήσεις και τότε θα διατεθεί πάλι χρήμα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτό, αυτή είναι η μέθοδος. Οι ανάγκες του Μαρτίου και για τα ομόλογα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν το δικαίωμα στα ισοζυγιά τους να έχουν ε, τέτοια δυνατότητα. Αυτό λοιπόν ισχύει. Δεν μπορεί απλώς να το ομόλογα. Και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για λόγου σταθερότητα να το δεχτεί αυτό για τις τράπεζες. Τις έχει προστατεύσει και αυτό νομίζω ότι είναι μια σοφή απόφαση. Και η τελευταία σα ερώτηση για δύο συγκεκριμένα μέτρα δεν τα γνωρίζω, δεν τα έχω εκτιμήσει εγώ, οπότε δεν μπορώ να αντιδράσω σε συγκεκριμένε προτάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε για το έργο κύριο Σκυρτσόφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. είμαι μερικούς μήνες ε, ευρωβουλευτής, αλλά είμαι 35 χρόνια οικονομικός συντάκτης και νομίζω ότι η προηγούμενη ιδιότητά μου με βοηθάει να καταλαβαίνω καλύτερα τα πράγματα γιατί εδώ χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε μια διπλωματική γλώσσα η οποία πολλές φορές δεν έχει σημασία. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει γίνει ένα σοβαρό λάθος στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης από την πλευρά του Eurogroup και νομίζω ότι η απάντηση που έδωσε ο κύριος Ντάισελμπλουμ στην ερώτηση της κυρίας Καηλή το επιβεβαιώνει. Δηλαδή δεν υπάρχει χρηματοδότηση επαρκής για το ελληνικό δημόσιο για τους επόμενους τέσσερις μήνες. Ε, για παράδειγμα, διαβάζω στον οικονομικό τύπο τον ελληνικό, χρειαζόμαστε 7,5 δισεκατομμύρια το Μάρτιο για τους πιστωτές μας, για το βραχυπρόθεσμο δανεισμό, για τα T-bills που δεν πρόκειται να επανεκδοθούν. Κανείς δεν ξέρει πώς θα καλυφθεί αυτό το πράγμα για να υπάρξει βέβαια κλίμα εμπιστοσύνης. Και υπάρχει βέβαια και ε, μια ανάλογη πορεία από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα πέφτουν με ρυθμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ το μήνα. 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήταν οι απώλειες τον Ιανουάριο, 1,2 δισεκατομμύρια εμφανίζονται οι απώλειες το Φεβρουάριο και η συζήτηση από την κυβέρνηση, τη νέα κυβέρνηση, είναι θα κάνει ένα πρόγραμμα, θα κυνηγήσει τους πλούσιους και θα φέρει στο μέλλον 5 έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόσθετα έσοδα. Μα με το ρυθμό που πηγαίνουν τα πράγματα θα έχει χάσει 10, 12, 14 δισεκατομμύρια έσοδα μέσα σε ένα χρόνο από την κατάρρευση του συστήματος. Επομένως έχουμε ένα έλλειμμα χρηματοδότησης από την πλευρά του Eurogroup που κάτι πρέπει να γίνει για να καλυφθεί. Έχουμε ένα ε, τεράστιο έλλειμμα εσόδων από την πλευρά της νέα κυβέρνηση που δεν γίνεται τίποτα για να καλυφθεί και συζητάμε τώρα και λέμε ότι εντάξει ελέγχεται η ελληνική κρίση για να διαπιστώσουμε σε ένα μήνα ότι όλα είναι εκτό ελέγχου. Ποια είναι η άποψή σας. I was waiting for the question. Περίμενα το ερώτημα ουσιαστικά. Τέλος πάντων, στο τέλος το άκουσα. Ήρθε και το ερώτημα. Θα δούμε τι θα γίνει τους επόμενους ε, δύο μήνες. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συνομιλήσει με τους θεσμούς ε, ε, δεν ξέρω ακριβώς ε, η κατάσταση που λέτε την οξία σε ό,τι αφορά την ταμιακή ροή, δεν ξέρω σε πόσο βαθμό σοβαρή και πόσο σοβαρή για την ελληνική κυβέρνηση. Το σημαντικό είναι το πρόγραμμα, η συμφωνία, η σύμβαση ε, είναι σε τροχιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξαναξεκινάμε και γι' αυτό θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πρόοδο. Και αν υπάρχει πρόοδο, τότε μπορούν να λάβουν χώρα και εκταμιεύσει. Έτσι έγινε με την προηγούμενη κυβέρνηση και έτσι θα γίνει και με την νυν κυβέρνηση. Το απλό γεγονό ότι υπάρχουν χρηματοδοτικέ ανάγκε δεν σημαίνει ότι θα αναστραφεί ε, αυτή η σειρά, θα αντιστραφεί ε, η τάξη αυτή. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο. Υπερβάν Μπερέ από του Σοσιαλδημοκράτε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, για την Ελλάδα, δεν έχετε την εντύπωση ότι μια από τι δυσκολίε οφείλεται εν μέρη στο ότι η απερχόμενη κυβέρνηση είχε ουσιαστικά επιθυμία να εξασφαλίσει την επανακλογή της Αφήνοντα την επανεξέταση του προγράμματο μέχρι το τέλο Φεβρουαρίου για τη νέα κυβέρνηση, αυτό πίεσε του πάντε και δυσκόλεψε τι συνθήκε των διαπραγματεύσεων. Έπειτα για τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει, είπατε και ο ίδιο ότι είχαν αντίκτυπο στη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών. Δεν συμμερίζεστε την άποψη ότι πολλέ από τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει ε, έχουν αποπληθωριστικό αντίκτυπο. Δηλαδή, ο ρυθμό των διαστατικών μεταρρυθμίσεων είναι κάτι που πρέπει να μα απασχολήσει. Ε, αλλά να το δούμε πιο ήρεμα, με περισσότερο χρόνο και όχι μόνο να κοιτάζουμε να πιέσουμε για την ε, μεταρρύθμιση των συνταξιδοτικών ε, συστημάτων. Εδώ τώρα απευθύνουμε σε ένα από τους τεσσάρους προέδρους, τεσσάρους, τέσσερις συν ένας, που την σύνοδο του Eurogroup στις 24 Οκτωβρίου ε, του περασμένου έτους συζήτησαν την παράταση της περασμένης θητείας. Οι εργασίες σας ξεκίνησαν ε, τη εγκαίρως αλλά δεν είχαν ομαλό ρυθμό. Ποια ήταν η άποψή σας για το αναλυτικό σημείωμα που είχε προβλέψει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής διότι η εντολή που, είχαν από το, η εντολή που είχε από το Eurogroup αναφερόταν στην αλληλεγγύη και την σύγκληση. Και αυτό το αναλυτικό σημείωμα αναφερόταν ακριβώς στην σύγκληση στο τέλος, στην τελευταία σελίδα του εγγράφου. στον όρο αυτό και μάλλον νομίζω με αρνητική χρειά. Και επίσης νομίζω ότι το σημείωμα αυτό ε, παραβλέπει τελείως όσα έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 όταν ανέλησε τις συνθήκες της Ευρωζώνης και το πόσο μεγάλες αποκλήσεις υπάρχουν. Μίλησα για τους πολλαπλασιαστές, για τον αποπληθωρισμό, για τις επιπτώσεις spillover. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα εν τέλει και συμμερίζεστε αυτή τη διάγνωση που ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έθεσε επιτάπητος. Um, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Το πρώτο ερώτημα ήταν κατά πόσο ε, η ατζέντα των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα χρειάζεται ή όχι περισσότερο χρόνο. Το ερώτημα είναι πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Κυρία Μπέρε, το ερώτημά μου είναι η αξιολόγηση του προγράμματος αναβλήθηκε λόγω των εκλογών στην Ελλάδα για τα τέλη Φεβρουαρίου, που σημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση δέχεται πλέον πολύ έντονες πιέσεις ε, σε αυτή την περίοδο από τις εκλογές μέχρι την νέα αυτή αξιολόγηση. Νομίζω όμως ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό το είχε ορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση και προηγούμενη κομισιόν με την ιδέα ότι θα συνεχίσουν όλα κατά τον ίδιο τρόπο. Κύριε Σντάιζεβλουμ, όχι, όχι. Ο λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα παρατάθηκε μόνο για λίγους μήνες ε, έχει να κάνει με διάφορες εθνικές εκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Έτσι λαμβάνουμε κάποιες φορές αποφάσεις. Μας είπε δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, έχουμε προεδρικές εκλογές πρόωρα. Προσπάθησαν τέλο πάντων, δεν έγινε αυτό, να εκλεγεί ο πρόεδρο και είχαμε πει ότι δύο μήνε μα φτάνουν, είχαν πει στην ελληνική κυβέρνηση. Με την ε, παράταση τώρα, ε, η κυβέρνηση έχει έξτρα χρόνο για να επεξεργαστεί τα σχέδιά τη, ε, τα οποία έπειτα, εφόσον ε, θεωρηθούν ότι συμβάλλουν ε, στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. Σωστά λοιπόν λέτε ότι το χρονοδιάγραμμα ήταν πάρα πολύ σύντομο για τη νέα κυβέρνηση, για να μπορέσει η νέα κυβέρνηση να συζητήσει τις μελλοντικέ ε, ρυθμίσεις, τους μελλοντικού διακανονισμούς και γι' αυτό προσπαθούμε τώρα να βρούμε το χρόνο και γι' αυτό δίνουμε αυτόν τον έξτρα χρόνο, βέβαια με κάποιους περιορισμούς, μέσα σε κάποια όρια. So second... Το δεύτερο ερώτημά σας τώρα αφορούσε το αναλυτικό σημείωμα του Προέδρου Γιούγκερ το οποίο ε, υποβλήθηκε εκ μέρους και των τριών άλλων προέδρων. Με ρωτάτε αν το υποστηρίζω και αν συμφωνώ με την ανάλυση του. Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα είναι ναι. Το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τώρα τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης ε, ε, δεν νομίζω ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Ήταν να συντάξει τον Ιούνιο με την έκθεση και θα πρέπει να προηγηθεί συζήτηση και μεταξύ των τεσσάρων πρόεδρων αλλά και με το Κοινοβούλιο, με τα κράτη-μέλη. Άρα ο πρόεδρος Γιούγκερ νομίζω ότι είναι αποφασισμένος να βάλει όλους αυτούς τους ε, φορείς να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν ε, μαζί του. Και θα περιμένουμε για τον Ιούνιο αυτή την έκθεση. Αυτό ήταν ένα απλά ένα αναλυτικό σημείωμα που έλδειχνε πώς στάσαμε σε αυτή την κρίση, τι πρέπει να κάνουμε, τι κάναμε μέχρι τώρα. Αν με την κρίση καταφέραμε τέλος πάντων να ενισχυθούμε, να οργανωθούμε, η απάντηση είναι ναι, αν αρκούν αυτά, η απάντηση είναι όχι. Θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Αυτό όμως είναι το χρονοδιάγραμμα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Για το ΕΛΚ. Τόμ Βαντεν Καντελάρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να σα απευθυνθώ στα Ολλανδικά, εφόσον είναι δυνατόν. Ακούσαμε πάρα πολλά για την Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το μέλλον, το μέλλον του δικού σας ρόλου, αλλά και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για το δικό σα ρόλο, η Ελλάδα Αναφέρατε ποια είναι τα συμφέροντα του Eurogroup και ο ρόλος αυτός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι ο συνδυασμός με τις ευρωπαϊκές υπουργικές θέσεις μου φαίνεται ότι δεν είναι ιδανικός. Σε καμία περίπτωση, μήπως ήταν καλύτερο να κοιτάξουμε μια μόνιμη προεδρία, όπως είπε ότι εκπρόσωπος αντιπρόεδρος, όπου ο επίτροπος που θα είναι πρόεδρος, γιατί, που θα είναι υπεύθυνος για θέματα νομισματικής ένωσης ε, θα πρέπει να έχει μόνιμη θέση στο Eurogroup. Για το ευρωπαϊκό εξάμεινο τώρα. Είναι πολύ σημαντικό το εργαλείο. Το πιο σημαντικό για την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής ε, Νομισματικής Ένωσης. Αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συστάσεων του εξαμήνου και αυτών που κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσει για την ανάπτυξη και τι θέσει απασχόληση δεν εφαρμόζονται επαρκώ. Και έτσι υπάρχουν μακροοικονομικέ ανισορροπίε, οι οποίε και αυτέ με τη σειρά του διακυβεύουν την Ευρωζώνη. Στην παρούσα φάση διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πετύχει να γίνει πιο δυνατή αν απαλύνει αυτές τις μακροοικονομικές ανισότητες. Πώς μπορούμε λοιπόν να δράσουμε προληπτικά για το μέλλον και να φροντίσουμε να αυξηθεί ο ρόλος και η σημασία των συστάσεων του εξαμήνου. Για παράδειγμα, να υπάρχουν ε, συμβάσεις με τα κράτη-μέλη με τις οποίες θα δεσμεύονται να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με τη συνοδεία φυσικά μηχανισμών αλληλεγγύης ε, σε ό,τι αφορά δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει για το δικό μου, με το δικό μου ρόλο. Όχι προσωπικά φυσικά, αλλά με την προεδρία του Eurogroup. Έχετε δίκιο. Πρόκειται για ένα ρόλο διαμεσολαβητή, θεματοφύλακα των διαδικασιών στο Eurogroup. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, τα πράγματα ήταν δύσκολα και ήταν δύσκολο να το συνδυάσω αυτό με τα καθήκοντά μου στην πατρίδα μου. Τα κατάφερα ωστόσο. Αλλά φυσικά ήταν και αρκετά έκτακτη και κατεπήγουσα η κατάσταση στα δυόμιση, στα δύο χρόνια μάλλον που ασκώ τα καθήκοντα αυτά. Τέτοιου είδους ε, ε, ένταση έχουμε παρατηρήσει μία μόνο φορά και καταφέραμε να τα βγάλουμε πέρα και στις δύο περιπτώσεις. Για το μέλλον τώρα. Πιστεύω ότι το Eurogroup αποτελεί ένα άτυπο διακυβερνητικό μέρος συνάντηση των Υπουργών και θεωρώ ότι θα ήταν παράλογο υπό αυτήν την έννοια να προεδρεύει του, της συνεδρίασης αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και πλεονεκτήματα στο γεγονός ότι ένας υπουργό προεδρεύει του Eurogroup, γιατί και ο Υπουργό αντιμετωπίζει την ίδια πολιτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν και οι συναδελφοί του και μπορεί να καταλάβει καλύτερα τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, τη δυσκολία προώθηση των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Όπω ξέρετε, η συζήτησή μου λύγει το καλοκαίρι. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει άλλη μια στιγμή αξιολόγηση, αν θέλετε για το εξάμεινο τώρα και τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ θεωρίας και πράξης. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η προώθηση μεταρρυθμίσεων πολιτικά έχει βάρος σε όλες τις χώρες και στην δική σας τη χώρα. Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις ε, που έχει συστήσει επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν περάσει ακόμα. Το ίδιο ισχύει και την δική μου χώρα. Εξαρτάται από την αποφασιστικότητα των εθνικών ε, πολιτικών. Των πολιτικών να πείσουν τους εκλογείς τους να τους επιτρέψουν τις μεταρρυθμίσεις αυτές. στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισοτήτων υπάρχουν δυνατότητες για να κλιμακώσει τις δράσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να σχέσει πιο πολύ πίεση. Δεν το έχει πράξει ποτέ ως τώρα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις το να υπάρχουν κυρώσεις, να υπάρχει δυνατότητα κυρώσεων, να υπάρχει δυνατότητα άσκησης πίεσης στα κράτη-μέλη. Αν τα κράτη-μέλη πραγματικά δεν αντιδρούν και δεν ε, αντιμετωπίζουν τις ε, κορυφαίες ανισότητε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να δράσει. Και αυτό μπορεί να γίνει και φέτος. Τέλος, μιλήσατε για συμβάσεις. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια σύμβαση. Η σύμβαση είναι ότι από κοινού έχουμε την ευθύνη να αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τις μακροοικονομικές ανισότητες, ιδιαίτερα αν υπάρχει μεγάλος αντικτύπος διασυνοριακά στην Ευρωζώνη και όπως σας είπα έχει ρόλο να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει εργαλεία στη διάθεσή της για να ασκήσει πίεση στις χώρες, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να ασκούμε πίεση και οι μεν στους δε. Αυτό γίνεται όλο και πιο πολύ στο Eurogroup, όπου οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν και φέρνουν ε, πραγματικά αντιμέτωπους τους συναδέλφους για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα θέματα στην εκάστοτε χώρα. Ευχαριστώ. Ο Πέτερ Σίμον, ο αντιπρόεδρο μα. Κύριε Ντάισελμπλουμ, το στυλ τη νέα ελληνική κυβέρνηση έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς ε, ανθρώπου. ιδιαίτερα στη χώρα μου. Παράλληλα, βλέπω σε πάρα πολλέ εκδηλώσει στη χώρα ότι ο κόσμο καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι ο ελληνικό λαό δεν θέλει να αποδεχτεί πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε και ο ίδιο ο λαός να αποδεχτεί. Όπως για παράδειγμα η Γερμανία. Ε, Ιδιωτικοποίηση, υγειονομικό σύστημα, συντάξει. Τα τονίζω αυτά γιατί, γιατί καλωσορίζω το γεγονός ότι αναφέρθηκε η λέξη ευελεξία από το στόμα σα. Για να αλλάξουμε κάποια μέτρα αν ε, οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Το ίδιο αποτέλεσμα α με άλλα μέτρα, αλλά σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Πολύ γρήγορα μπορεί να πετύχουμε αποτελέσματα να περικόψουμε συντάξει, αν ιδιωτικοποιήσουμε πιο δύσκολα και πιο αργά, αλλά με το ίδιο τελικά αποτέλεσμα θα πετύχουμε με φορολογική μεταρρύθμιση. Η ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει με το χρονικό ορίζοντα. Εσείς προσωπικά, ως πρόεδρος του Eurogroup, είστε αντιτεθειμένος στα πλαίσια της ευελιξίας την οποία και επικροτείτε, αν οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Να διαπραγματευτείτε με την Ελλάδα και να μιλήσετε για θέματα χρονικού ορίζοντα, αν είναι σαφές ότι το ίδιο αποτέλεσμα τελικά θα επιτευχθεί. Η απάντηση. Ο βασικός μου στόχος θα είναι ο εξής. Να υπάρξει βιώσιμη συμφωνία με την Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει ότι τα μέτρα τα οποία θα συμφωνήσουμε μπορούν ρεαλιστικά να εφαρμοστούν στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο. Κάποια από τα μέτρα τα οποία έχει προτάξει η, Ευρωπαϊκή, η ελληνική κυβέρνηση, που υποστηρίζω, όπως για παράδειγμα ένα υγιές φορολογικό σύστημα, θα πάρουν χρόνο. Πολλά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη και την τεχνική αρρωγή της Γερμανίας, ε, της Ολλανδίας και άλλες χώρες ε, συνέδραμαν για να υπάρξουν καλύτερε φορολογικέ υπηρεσίε στην Ελλάδα, αλλά παίρνει χρόνο. Και το θέμα δεν είναι μόνο να περάσει νομοθεσία στο Κοινοβούλιο. Ένα από τα πράγματα που μάθαμε από τα προγράμματα του παρελθόντος είναι το εξή. Το ότι να περνάνε ε, νόμοι από τη Βουλή είναι τελείω διαφορετικό πράγμα από το τι συμβαίνει με την πραγματικότητα. Το τι γίνεται στην όλη διαδικασία εφαρμογής όλα παίρνουν χρόνο. Θα πρέπει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα για την Ελλάδα ρεαλιστικό που θα καταστήσει πιο στεναρό τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Ελλάδας αλλά και που θα είναι ρεαλιστικό σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας ωστόσο τώρα. Κάποιοι από τους στόχους που έχουμε θα πάρουν πιο πολύ χρόνο. Αυτή είναι η ρεαλιστική αξιολόγησή μου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Follow-up. Επερώτηση. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, επιτρέψτε στο σημείο αυτό να κάνω μια επερώτηση. Η ανάλυση η οποία κάνατε επί της ουσίας καταδεικνύει ότι ναι υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να πετύχουμε στο χρονικό ορίζοντα. Αν συμφωνούμε όμως ότι η εφαρμογή μιας μεταρρυθμίσης στο φορολογικό σύστημα τελικά θα οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα, μπορούμε να δείξουμε προθυμία να συζητήσουμε και το χρονικό ορίζοντα για να περάσουν πραγματικά βιώσιμες μεταρρυθμίσεις. Η επωνομαζόμενη Τρόικα κατάφερε στο παρελθόν να πετύχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θεωρούνταν δύσκολα. Μπορούμε να καταφέρουμε να πετύχουμε σε ένα άλλο δύσκολο σημείο στο να πούμε στους λαούς της Ευρώπης ότι σε κάποια θέματα χρειαζόμαστε άλλο χρονικό ορίζοντα για να περάσουν βιώσιμα κάποιες αλλαγές στην καθημερινή ζωή. Ενδεχομένω η φορολογική μεταρρύθμιση να βοηθήσει σημαντικά στην επίλυση χρηματοπιστωτικών προβλήματων. Πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχει τεράστιο δυναμικό στην Ευρώπη. Θα πάρει πολύ χρόνο. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε στο μεταξύ, σε ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Αν επιτρέψουμε στον, ευρωπαϊκό, στον ελληνικό προπολογισμό να ξεφύγει τα επόμενα χρόνια και η βιωσιμότητα του χρέους επίσης θα ξεφύγει. Θα πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποδεχτούμε να μην συμβεί τίποτα πρόθεσμα και να ξεφύγει τελείως ο προϋπολογισμός ενώ προσπαθούμε να επαναδιοργανώσουμε και να επανειδρύσουμε ένα υγιές φορολογικό σύστημα, ένα ε, ε, εύρυθμα λειτουργικό σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν και ο προπολογισμό και το χρέο να παραμείνουν υπό έλεγχο. Πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να επιλέξουμε ή το ένα ή το άλλο. Και τα δύο θα πρέπει να το κάνουμε. Και μεταρρυθμίσει και χρέο και προπολογισμό. Ιδάλω θα χρειαστούν περαιτέρω χρέωση και θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του ελληνικού χρέου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις της βάσης του προγράμματος. Να κατανοήσουμε ότι εντός του Eurogroup υπάρχει σαφώς η άποψη για το αν είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα και σε ποια σκέλη του, τι πέτυχε και τι όχι, ή το μόνο πρόβλημα είναι η έλλειψη επίτευξης πρόοδο από τους Έλληνες. Um... Βεβαίω η απουσία επιτυχών αποτελεσμάτων είναι μέρος του προβλήματος, αλλά ένα άλλο μέρος είναι ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές. Ένα άλλο κομμάτι της απάντησης είναι ότι ορισμένα ζητήματα που μόλις συζητήσαμε απαιτούν πολύ χρόνο. Δεν είναι μόνο το θέμα της πρόθεσης νομοθεσίας ε, δεν αρκεί ε, να περνάνε τα σωστά νομοθετήματα. Υπάρχει και η μακρά και πολύ δύσκολη και πληκτική φάση της υλοποίησης, επίσης η ανάληψη καθηκόντων από νέα κυβέρνηση. Με όλους αυτούς τους νέους παράγοντες η απάντηση είναι η σύνθεση όλων αυτών. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως είχα πει και στα τέλη της περασμένης χρονιάς, το πρόγραμμα πρώτη φορά έφερα αποτελέσματα ω προ την οικονομική ανάπτυξη και τι αποδόσει, αποτελέσματα την περασμένη χρονιά. Ήδη τα φορολογικά εισοδήματα άρχισαν να αυξάνονται πέρυσι στο τέλο τη χρονιά και τώρα ξαφνικά έπεσαν πάλι. Η φιλοδοξία μου είναι, και ελπίζω να επιτύχει σε αυτό η ελληνική κυβέρνηση, να συνεχίσει από εκεί που ήταν η Ελλάδα πριν από ένα εξάμεινο, όταν είχε επανέλθει ανάπτυξη, τα φορολογικά εισοδήματα αυξάνονταν και πρώτη φορά δημιουργόταν θέσει μετά από πολλά χρόνια. Αυτό θα θέλαμε να ξαναρχίσει και να συνεχιστεί και να το στηρίξουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε το χρόνο που είχαμε για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρον, φοβερά επικοδομητική συζήτηση. Μπορούμε να καλωσορίσουμε και να χαρούμε για την αισιοδοξία αυτή, τη θετική ε, προσπάθεια του Eurogroup και του Προέδρου του που προσπαθούν να έχουν μια επιτυχή ε, κατάληξη σε αυτές τις δύσκολες συνομιλίες. Το ίδιο το σύστημα της νομικής ένωσης ε, τέθηκε επιτάπητος και έπρεπε να βρεθεί η σωστή διάρθρωση της αρχής της ε, νόμιμης δημοκρατίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος και μιας κυβέρνησης που μπορεί να, αποφα... να λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις, κυρίαρχες αποφάσεις, αλλά και τις διεθνείς δεσμεύσεις που επηρεάζουν και άλλες χώρες. Εδώ λοιπόν οι μελλοντικέ θεσμικέ εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και βεβαίως αναμένουμε την επόμενη παρουσίαση του Προέδρου, ε, θέλουμε να δούμε κατά πόσον μπορεί να υπάρξει κοινοτικοποίηση της δημοσιονομικής στήριξης των κρατών μελών. Αυτό μεσοπρόθεσμα καλό να το σκεφτούμε εάν θέλουμε να συμφιλειώσουμε καλύτερα τα δικαιώματα των εθνικών δημοκρατικών κρατών αλλά και την ανάληψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν μιλάμε για ε, αλληλένδετα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και καλή τύχη για την υπόλοιπη δουλειά σας. Dear colleagues, we have Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι και ό,τι πρέπει γιατί αύριο ψηφίζουμε σχετικά για την έκθεση Ροζάτη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ε, παρακαλώ. Παρακαλώ καθίστε. Yeah. Thank you. Thank you very Thank much. You. Okay. See you next time. Right. Bye. As you know, όπως θα ξέρετε, παραδοσιακώς η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την ετήσια, έκθεση, για την ετήσια έρευνα ανάπτυξης μας δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθούμε ως προς τις οικονομικές εξελίξεις, τη στρατηγική τριών πυλώνων που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια σημαντική στιγμή για το ρόλο που έχουμε αναλάβει και εμείς στα πλαίσια της δημοσιονομικής ε, Ένωσης στην Ευρώπη. Να δώσω, αύριο θα ψηφίσουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε να δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντάριος Ροζάτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω ότι η έκθεσή μου δεν είναι τόσο συναρπαστική όσο τα προηγούμενα σημεία της ημερής διάταξης. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε το σοου με το πρόγραμμα δηλαδή. Να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές που εργάστηκαν σκληρά για να καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα ήταν αποδεκτή για την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Είχαμε επικοδομητικές συζητήσεις και η εντύπωση μου είναι ότι όλοι εργαστήκαμε για ένα κοινό στόχο μια έκθεση που θα αποτελέσει μια πραγματική συνεισφορά για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να υπάρχει προστιθέμενη αξία στη διαδικασία καθορισμού πολιτικών προτεραιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτόν τον κύκλο των εθνικών οικονομικών πολιτικών εντός του Ευρωπαϊκού Ξαμήνου. Η άποψή μου είναι ότι εν τέλει έχουμε καταλήξει σε λογικέ συμβαστικέ λύσει. Δεν συμφωνήσαμε σε όλα φυσικά. Υπάρχουν ακόμα διαφωνίε σε πολλά θέματα. Αλλά η εντύπωσή μου είναι ότι στο πνεύμα καλή συνεργασία, ώστε να έχουμε κάτι χειροπιαστό, συγκεκριμένο και θετικό, καταφέραμε σε πολύ σημαντικά τμήματα τη έκθεση να πετύχουμε συμφωνίε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε αλλά θέλω να ακούσω τις απόψεις των εκπροσώπων άλλων πολιτικών ομάδων για το σχέδιο. Αυτό που προέχει και ήθελα να προσκαλέσω τους συναδέλφους να θυμούνται ότι ο βασικός στόχος της έκθεσης είναι ότι όλοι θέλουμε η Ευρώπη να πάρει το δρόμο της γρήγορης ανάπτυξης με ενίσχυση του ανταγωνισμού, με πιο καλοπληρωμένες δουλειές και λιγότερη φτώχεια. Αυτός είναι ο απότερος στόχος που θα πρέπει όλοι να συμμεριστούμε. Να ακούσω και να, να πω τώρα ότι είμαι ανοιχτό στα σχόλια των υπολοιπών συναδέλφων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον σκιώδη συγκητή από την Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ομάδα, τον κύριο Αλφερτ Σάντο. Ο Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ροζάτη γιατί έλαβε πολύ ε, ευφύς πρωτοβουλίε ε, και συνεισέφεραν ε, και οι άλλοι σκιώδεις. Βέβαια, δύο διαφορετικές εκτιμήσεις τη οικονομική πραγματικότητας βλέπουμε. Από τη μία, κάποια από εμά θεωρούμε ότι η δημοσιονομική εξυγίαση και οι διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητε. Και από την άλλη πλευρά, κάποιοι άλλοι πιστεύουν, και είμαι ένα από αυτού ότι χρειάζεται να δοθεί ε, μια δημοσιονομική τόνωση. στι τελευταίε εβδομάδες Είδαμε ότι είναι πολύ κοντά στην αλήθεια αυτή η άποψη και χρειάζονται κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Θα συνεννοηθούμε με τον κύριο Ροζάτη για τα πιο πολλά μία εξαίρεση υπάρχει. Προσπαθούμε να εστιάζουμε στα πραγματικά στοιχεία. Δεν σημαίνει βέβαια ότι διάφορες προτάσεις ε, εξαλλήλω αποκλείονται πρέπει να δούμε κάποιους ορισμούς όπως διαστατικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης δεν θα πρέπει το κοινωνικό μοντέλο να διαφραθεί, να απαλληφθεί. Κατώτατη μισθή, συντάξεις, ε, επιδόματα είναι σημαντικά. Δεν πρέπει να μειωθούν. Βέβαια, πρέπει να καταργηθούν τα μονοπόλια, πρέπει να είναι σωστή υπάρχει των υπηρεσιών. Πρέπει να μειωθεί η κρατική γραφειοκρατία, να εξορθολογιστούν οι πρακτικές των δημοσίων διαγωνισμών και προμηθειών. Τέτοιες δραστικές μεταρρυθμίσεις ε, θα τις στηρίξουμε. Υπάρχει οριστία σε κάποια πράγματα. Η οικονομική και η κοινωνική σύγκληση είναι σημαντικό στοιχείο και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα δούμε επίση πώ θα διαμορφώνονται οι εθνικέ πολιτικέ και πώς συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών. Δεν έχουμε ένα προοδευτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση εθνικών περιφερειακών ε, διαφορών και ανισοτήτων. Θέλουμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο οικονομική διακυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να θεραπεύσουμε τι διαφορετικέ ανισότητε και αδυναμίε τη Ένωση. μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά λίγο πιο αργά. The dogma of fiscal consolidation has become... Η δημοσιονομική εξυγίανση είναι μια πολιτική που δεν έδωσε λαμπρά αποτελέσματα. Η τροποποιηθής έκθεση δείχνει επίσης και το ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Πρέπει απλά να δούμε αν το ποτήρι, το ποτήρι να το δούμε ως μισογεμάτο και όχι ως μισοάδιο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν βελτιωθεί εξίσου, όπως η ΣΥΠΑ ή αλλού. Δεν είναι σαφής η απάντηση γιατί δεν έγινε αυτό. μπορούμε να πετύχουμε. Το έδειξε η κυβέρνηση της Ελλάδας δημοκρατικές αλλαγές και μπορεί να κινητοποιηθούν και άλλοι λαοί μετά από αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Το θέμα που θα μπορούσε να προκύψει μεταξύ άλλων της Ευρώπης είναι ποιος ωφελείται από όλα αυτά. Αλλά αυτό θα μπορούσε να διχάσει τον κόσμο να χωρίσει το βορρά από τον νότο, την Ανατολή από τη Δύση. Το θέμα είναι να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή και συνεκτικότητα. Δεν είμαι πεπισμένος ότι τα σημεία τα οποία σας ανέφερα είναι μακριά από τους στόχους όπως μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν. Και αν το θεωρήσουν, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Παραλαμβάνω υπάρχουν κοινωνικέ και οικονομικές ανισότητες, πάντοτε υπήρχαν φαίνεται να βαθαίνουν. Ο στόχο μας είναι πολιτικός κυρίω. Όπου και αν ανήκουμε θα πρέπει να δούμε αυτό το έγγραφο που θα ψηφίσουμε αύριο για αυτή την ετήσια έρευνα και επισκόπηση για την ανάπτυξη. Και να αναφέρω τώρα τις συμβιβαστικές για τις ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που δεν συμφωνήσαμε αν περάσει η τροπολογία θα καταψηφίσουμε σοσιαλδημοκρατική ομάδα και συγκεκριμένα θα σας το αφήσω να το ακούσετε. Private investments have increased because of stronger market confidence and lower interest rates, while the governments have tried to stimulate the economy through deficits and increase public spending, investments have fallen and unemployment risen. End of quote. Αν περάσει αυτό το σημείο, εμείς θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Τέρχο από τους συντηρητικού και Μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε εισηγητά, συνάδελφοι, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρο τη. Είναι πολύ καλή έκθεση από πολλέ σκοπιές. Πιστεύουμε ότι ο εισηγητή ήταν πολύ επιτυχής στον τρόπο που ανέλησε την οικονομική κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, πολλέ από τι λύσει που προτάθηκαν στην έκθεση είναι ρεαλιστικές και μπορέσαμε να εντοπίσουμε πολλά από τα προβλήματα που, εντοπί, που προκαλούν τις οικονομικές δυσχέρειες στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, όπως συγκεκριτής πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη κρατήσει τις υποσχέσεις της για την δημιουργία της ενίας αγοράς, ιδίως για, την υπηρεσία, για τις υπηρεσίες και την ψηφιακή οικονομία. Όμως η έκθεση αυτή και πάλι έχει κάποια θεμελιώδη, κάποια προβλήματα επί τη ουσία που μας κάνουν πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να τη στηρίξουμε. Πλήρως τουλάχιστον. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι παρόλο που το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μπορεί να παράσχει επαρκή συμβουλευτικό ρόλο προ τα κράτη-μέλη, ο ρόλο είναι καθαρό συμβουλευτικό και δεν θα πρέπει να υπονομεύει τι εξουσίε των κρατών μελών υπό οποιαδήποτε μορφή. Γι' αυτό δεν μπορούμε να στηρίξουμε καμία περίπτωση επιβολής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και είμαστε ιδιαίτερα ε, επιφυλακτικοί για το να γίνουν οι συστάσεις δεσμευτικές για τα κράτη-μέλη. Όμως μεγάλο πρόβλημα είναι και η θεσμοθέτηση της Τρόικας διότι δεν πιστεύουμε ότι με την έλλειψη δημοκρατικής λογοδοσίας της Τρόικας μπορούμε να έχουμε την κατάλληλη νομική υπόσταση για να συνδυαστεί με τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. Πιστεύουμε η Τρόικα δεν πρέπει να υπάρξει καν στο μέλλον. Θα πρέπει να καταργηθεί. Αυτέ οι λεπτομέρειε λοιπόν έχουν καταστήσει πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτήν την συνολικά πολύ καλή και καλά συντεταγμένη έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τόρβαλτς για του ελευθέρους. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Ροζάτη για τη δουλειά που έκανε. Δεν ήταν ε, σε καμία περίπτωση απλό το έργο του, γιατί όπως ξέρουμε, σε τέτοιου είδους συζητήσει. ακούγονται όλες οι πτυχές του πολιτικού και ιδεολογικού φάσματος στην Ευρώπη. Ένας μικρό κοσμός της ε, συζήτησης που διεξαγάγεται και στο εξωτερικό του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι οι συμβιβασμοί ωστόσο είναι αρκετά ισορροπημένοι. Έχουμε μια έκθεση μπροστά μας που ακολουθεί την προηγούμενη γραμμή του προηγούμενη, της προηγούμενης έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η έκθεση λοιπόν αυτή, αν εγκριθεί σήμερα και μετά από την Ολομέλεια, νομίζω ότι θα εξυπηρετήσει. Θα είναι μια καλή βάση για τη συζήτηση για περισσότερη ανάπτυξη και οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή και μετά ασφαλώς. Με όλα τα αυτά, ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα ακολουθήσουν τις συστάσεις της έκθεσης, ακόμα και αν δεν δεσμεύονται με κανέναν τρόπο από μια τέτοια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε ιδεολογικός και πολιτικός πώς εξελίσσεται η συζήτηση. Νομίζω ότι έχουμε μία περίπτωση σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για την Ελλάδα και στο ιστορικό της Ελλάδας Πολλές από τις συζητήσεις ε, που γίνονται από την έκθεση της Τρόικας και από άλλες εκθέσεις και μετά εστιάζονται σε ευσεβείς πόθους. Ευσεβείς πόθους που δεν μας βοηθούν απαραίτητα σε κάθε φάση. Νομίζω λοιπόν ότι ο συνάδελφος Ροζάτη είχε πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά προκειμένου να συνενώσει όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και τώρα λέει ο Πρόεδρος για την ΚΟΕ. Το λόγο έχει ο Μιγγέλ Βιέγκας. Ευχαριστώ. Ως προς την έκθεση αυτή, να πω ότι θέλουμε να πετύχουμε να συμπεριληφθούν κάποιες από τις δικές μας παρατηρήσεις που αντακοτοπίζουν τις δικές μας απόψεις επί του θέματος, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη βαθιά μας διαφωνία με όλη αυτή τη διαδικασία και ιδίως τους λόγους που ουσιαστικά είναι και αίτια για την ε, οικονομική ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η κρίση αυτή είναι καρπός της ε, διαδικασίας ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς, της ε, υποταγής της ε, οικονομίας, της χρηματαγορές και της χρηματοπιστωτικές ανάγκες και το ίδιο και των πολιτικών αποφάσεων. Έτσι λοιπόν οι κεντρικοί θεσμοί ε, ουσιαστικά οδηγούν σε ναυάγιο την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Με την ευελιξία στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, με την αιμονία αυτή στη δημοσιονομική αυστηρότητα, με ε, ε, με το πρόγραμμα επενδύσεων και την πρόταση αυτή που προτείνει τις εταιρικές σχέσεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα με κόστος που καλύπτεται από το δημόσιο και κέρδη που πηγαίνουν τελικά στον ιδιωτικό τομέα όπως όλοι γνωρίζουν. Δεν πιστεύουμε ότι αυτές είναι οι λύσεις για τα προβλήματά μας. Πεποίθησή μας είναι να κοιτάξουμε τι γίνεται ε, ε, στην πραγματικότητα, δηλαδή ανεμική ε, ζήτηση σε ύφεση και σε πτώση ε, ανάπτυξη, χρέη, υπέρμετρα, λόγω των πολιτικών που ζητά να εφαρμοστούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το σημείο αφετηρίας που θα πρέπει να μας οδηγήσει να αναλάβουμε νέα μέτρα, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και η κοινωνική Ευρώπη να βρεθεί στο κέντρο των οικονομικών πολιτικών. Thank you. Ευχαριστούμε. Για τους πρασίνους ο κύριος Ουρτασούν. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ροζάτη για τον καλό διάλογο και την καλή του διάθεση για να συζητήσουμε τα διάφορα ζητήματα της έκθεσης. Ούτως ή άλλως ε, υπάρχουν ε, διαφορές σίγουρα για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε και εκτιμούμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο που θα μας κάνει να μην στηρίξουμε την έκθεση, πάντως να τον ευχαριστήσουμε που έδειξε καλό πνεύμα διαλόγου. Αμφισβητούμε πολλά από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ω ομάδα συμφωνούμε βέβαια ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμό των οικονομικών πολιτικών ε, των ε, κρατών μελών και πολύ περισσότερο στους τόνους να υπάρξει, όμως η διακυβέρνηση θεώρησε, θεωρήθηκε ως εργαλείο για διαδικασίες εσωτερικής υποτίμησης σε κάποιες χώρες. Επλέγησαν ιδίω τα κράτη-μέρη που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν κοινωνικοί δείκτες ε, και δεν συμπεριλαμβάνονται κοινωνικοί εταίροι σε όλες τις διαδικασίες, όπως και άλλοι παράγοντες. Οι δημοσιονομικοί στόχοι παίρνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Υποτιμούνται οι στόχοι της στρατηγικής 2020 ε, Αυτά τα σημεία δείχνουν σοβαρέ ανεπάρκειε του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κατά την άποψή μα. Διαφωνούμε επίση με την προοπτική ετήσια μελέτη ανάπτυξη το 2015. Υπήρχαν προσδοκίε ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή παραδείγματο στι οικονομικές πολιτικές και από το κοκτέιλ καθοδικών μεταρρυθμίσεων και λιτότητα θα περνάγαμε στη στήριξη των επενδύσεων, τη ανάπτυξη και τι κοινωνικής πολιτικής. Δεν έγινε έτσι όμω. Το κείμενο χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια, δημιουργία απασχόληση, κοινωνικές, ε, μάλλον πολιτικέ κοινωνική ισότητα πάλι μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο θεμελιώδη στοιχεία που έχουν μείνει εκτός λοιπόν ε, και άλλα που δεν ε, θέλουμε να είχαν συμπεριληφθεί. Επίση, ό,τι αφορά τι διαδροτικέ μεταρρυθμίσει, πάλι είναι σε κεντρικό σημείο. Σίγουρα ε, συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη. Καλό αυτό. Συνολικά όμω, Ξεκολουθούμε να θεωρούμε ότι το κείμενο αυτό είναι συγκαταβατικό, συμφωνεί με τι πολιτικέ τη Κομισιόν, δεν έχει διδαχθεί από το παρελθόν και ούτε αντιμετωπίζει το κίνδυνο του αποπληθωρισμού, τι εσωτερικέ ανισορροπίε, ίδιο πληρωμών ε, και τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού τον προανέφερα. Έχουμε και το πρόβλημα τη ανεργία. Η μόνη συνταγή που προτείνεται εδώ είναι αυτή τη Κομισιόν, δηλαδή συγκράτηση των μισθών. Σε πολλέ χώρε, ιδίω στην περιφέρεια, γίνεται ήδη. Περικόπτονται δικαιώματα και μειώνονται τα επιδόματα προς τους ανέργους. Δεν γίνονται και πολλά για την ε, ανάπτυξη, ούτε ε, και πολλά για την καταπολέμηση των ισοτήτων. Και ολοκληρώνω. Το κείμενο και η αξιολόγηση, αυτή η προοπτική μελέτη, είναι μεροληπτικά κείμενα. Αντικατοπίζουν φιλελεύθερα δόγματα αυτών που κυβέρνουν την Ευρώπη δεν εκφράζονται πολλές κριτικές, είναι συγκαταβατικό το κείμενο. 12 φορές αναφέρεται διορθωτικές μεταρρυθμίσεις και λέγεται ότι τα προγράμματα προσαρμογής εστέφσαμε επιτυχία. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά. Παρά λοιπόν το ότι έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες έγιναν δεκτές οι λιγότερο πολιτικά λεπτές από αυτές και οι πιο σημαντικές δεν ελήφθησαν υπόψη σας λέω λοιπόν ότι θα καταψηφίσει η ομάδα μας την έκθεση. Παραλαμβάνω όμως ότι ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για το καλό πνεύμα και για τη διάθεση για διάλογο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρου του Σκιώδης εισηγητή του, της ομάδας μου, του κ. Βάιλη, που δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή εδώ και ζητά συγγνώμη. Και εμείς ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δουλειά του καθώς και τους δυο συζητητές, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το κείμενο, το τελικό κείμενο της έκθεσης. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τα διάφορα σημεία που δεν μας ικανοποιούν και όπου θα θέλαμε να δείξει μεγαλύτερο θάρρος και τόλμη το Κοινοβούλιο. Το πρώτο σημείο είναι το εξής. Κατά την άποψή μας η έκθεση αυτή δεν δει καμία επί της ουσίας συνεισφορά για την ε, επίσημη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Το κεντρικό σημείο που πρέπει να επικρίνουμε είναι ότι πολλοί αρέσουν στην έκθεση αυτή τα μέτρα λιτότητας που προτάθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης. Είναι σαφές ότι ήταν αποτυχέστατα τα μέτρα αυτά και όχι απλώς δεν βοήθησαν να ε, ε, ξεπεραστεί η κρίση, αλλά την ε, επιδίνωσαν σε πολλές χώρες. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν το σημείο αυτό είναι τελείως άσκοπο. Θα έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερη τόλμη και να επικρίνουμε τα μέτρα αυτά που υιοθετήθηκαν. Ένα άλλο σημείο όπου δεν συμφωνούμε είναι η υπεραισιόδοξη άποψη της έκθεσης αυτής για τις προβλέψεις της μελλοντική ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεδομένου του αντικτύπου που θα έχει το επενδυτικό πρόγραμμα όπως προτείνεται από την Επιτροπή Juncker. Κάθε χρόνο βλέπουμε και το δείχνει η ιστορία και η πρόσφατη εμπειρία μας ότι όποτε μιλάμε για ανάκαμψη, μια σχετική ανάπτυξη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως μετά τα τελικά στοιχεία διαψεύδουν τις ελπίδες και ξαναβρισκόμαστε σε κατάσταση οικονομικής τελμάτωσης. Και υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, ίσως καλό θα ήταν να υπήρχε αλλαγή ως προς το επενδυτικό πρόγραμμα. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε όπως προτείνεται να προσφέρει ουσιαστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι Γίνεται λόγος για πρόσθετες προσπάθειες από δημοσιονομικής πλευράς. Αυτό που συνέβη τα περασμένα χρόνια θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο. Και γίνεται πολλή λόγος για διαστατικές μεταρρυθμίσεις. Διαστατικές μεταρρυθμίσεις που ισοδυναμούν με περικοπές, με αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας, με αποδυνάμωση της δημόσιας κληρονομιάς, δεν ε, ωφελείται κανείς βραχυπρόθεσμα, αυτό που το ή άλλω αλλά οι διαστατικές μεταρρυθμίσεις ακριβώς μπορεί να είναι επιζήμιες για την οικονομική ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα. Και τέλος ένα σημείο για το οποίο διαρκώς δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή της ανισότητες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις μακροοικονομικές ανισότητες και κυρίως εντός Ευρωζώνης. Γίνεται πολύ λίγος λόγος για τις ανισότητες του current accounting και κυρίως για την περίπτωση της Γερμανίας. Η ομάδα μου στην Επιτροπή ΕΚΟΝ υπέβαλε ερώτημα για το πλεόνασμα των λογαριασμών της Γερμανίας που δεν σέβεται τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας ήδη από τις, από τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εντοπίσει τις σημαντικές μακροοικονομικές ανισότητες εντός Ευρωζώνης. Και υπ' αυτή την άποψη λοιπόν θα πρέπει να δούμε ε, εάν μπορούμε να δείξουμε περισσότερο θάρρος στο να εντοπίσουμε τα μακροοικονομικά προβλήματα εντός Ένωσης και να προτείνουμε μέτρα για να τα λύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα, catch the Ματ ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να πω και εγώ από δική μου πλευρά ότι δεν υπάρχει κανένας σκοπός να συζητάμε τις προτάσεις για την ετήσια ανάπτυξη αν το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι τόσο σεγαδιασμένο για την Ιρλανδία, τη χώρα μου, αναβαίνει ότι είναι η προμονωτική χώρα με ισότητα σε ό,τι αφορά την κατανομή εισοδημάτων και κατά πόσον τα απόλυτα ευρήματα γίνονται αποδεκτά. Φαίνεται ότι πρόκειται για θέμα ανισότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δυστυχώ, του τουλεχθέντο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να χρονοτρεβεί με τι μεταρρυθμίσει του 2 pac και του 6 pac σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο για τον δρόμο προς την χειριαρχία και την οικονομική ανεξαρτησία πιστεύει και το κομμού πιστεύει ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην ε, μείωση της φτώχειας και όχι να αποφεύγουμε τους εκάστοτε οικονομικού κύκλους, γιατί η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προέλθει από την αντιμετώπιση των ισοτήτων και της ενοτροπίας που οδήγησε στην οικονομική κρίση την οποία και αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο, Δεν βλέπω να ζητάει κανεί άλλο το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασία του ΚΑΣΔΙ. ω εκ τούτου μπορώ να δώσω το λόγο εκ νέου στον εισηγητή. Κατανοώ ότι υπάρχουν κάποια αιτήματα προς τον εισηγητή για να καταβάλει μια παραπάνω προσπάθεια για συμβιβασμό και πολύ θα ήθελα να ακούσω και τα δικά σας σχόλια από αυτού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους κοιούντες εισηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων για τις συζητήσεις που κάναμε για μία ανοιχτή και ειλικρινή στάση και τα ανοιχτά τους σχόλια. Όπως προείπα, φυσικά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα πάντα. Είναι πολιτικό το ζήτημα και υπάρχουν και ουσιαστικές διαφορές στην αξιολόγηση διαφορών πτυχών της οικονομικής κατάστασης σήμερα. Να αναφερθώ σε κανένα δύο σημεία όμως στην παρούσα χρονική συγκυρία. Καταρχάς, θα μπορούσα να συμφωνήσω με διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν, με διάφορες τροπολογίες που κατατέθηκαν από τις 268 στο σύνολο Ασφαλώς όμως δεν μπορώ να τις βάλω όλες στην ε, έκθεση, πολύ απλά γιατί θέλω να επικεντρωθώ στο πεδίο εφαρμογής της ετήσιας έκθεσης ανάπτυξης, που δεν αφορά την καταπολέμηση της στόχιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην Οικονομική Ένωση, αφορά κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα. Πρόκειται για ένα σημείο κίνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που σκοπό έχει να συντονίσει καλύτερα τις εθνικές πολιτικές και βασικά σε δύο επίπεδα, μακρό χρηματοπιστωτικό επίπεδο και στο επίπεδο διορθωτικών μεταρρυθμίσεων. Θέλω να αποφύγω να έχουμε μία έκθεση που θα μιλάει επί παντός επιστητού και η οποία εκ παραλλήλου ήταν τόσο γενικόλογη που τελικά δεν θα έχει καμία επικέντρωση, καμία στόχευση, γιατί ασφαλώς ο αντίκτυπος της έκθεσης αυτής στη διαδικασία συντονισμού των εθνικών πολιτικών θα είναι αμεληταίος. Προσπαθώ να πείσω τους συναδέλφους ότι η έκθεση δεν είναι μια έκθεση για τα πάντα. Ασφαλώς έχουμε τοποθετήσεις για πολλά άλλα ζητήματα. Άρα, τους καλώ να εξετάσουν την έκθεση αυτή ως τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα και συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για την ανάπτυξη που αποτελεί τη βάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και για τις συστάσεις αναχώρα. Δεν είμαστε σε θέση στην παρούσα φάση να καλύψουμε ασφαλώς όλα τα σημαντικά ζητήματα με μία έκθεση. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα το απόγευμα, δεν έχει λοιπόν τόσο πολύ χρόνο δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο μπροστά μα. Φυσικά είμαι ανοιχτό για συζητήσει και για αλλαγέ τελευταία στιγμή, ενδεχομένω που θα μα επιτρέψουν να έχουμε μεγαλύτερη πλειοψηφία που θα υποστηρίζει το έγγραφο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα να ολοκληρώσουμε τι συζητήσει μα Προσβλέπουμε στην ε, σημερινή ψηφοφορία, σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ και πέρασε τη συνεδρία σας.